Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Για να δούμε μπορούμε να κρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Επίσης πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 22ης και 23ης Μαρτίου αλλά και τη 21 η Μαρτίου. Εγκρίνονται αν δεν έχετε σχόλια. Μία μόνο ανακοίνωση. Έντεκα και 30 θα το γνωρίζετε ασφαλώς. Έχουμε κοινή επιτροπή υπό το άρθρο 55 του κανονισμού μαζί με την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων για, την, ε, για το θέμα των εκθέσεων αναχώρα. Έχει ήδη οργανωθεί η διαρρύθμιση της ε, αίθουσας. Αυτό εξηγεί και τις αλλαγές της θέσης σας. Και το ίδιο για το απόγευμα με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ψηφοφορία μετά τις 6 και 20. κατά εξουδιώτηση πράξη μετά την οδηγία για την αντιμετώπιση της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Θέματα προκαταρκτικά δεν έχουμε γιατί τα είχαμε καλύψει πριν και πάμε στα σημεία 5 έως 9, δεύτερη ανταλλαγή απόψεων στην τραπεζική δέσμη, άνευ περαιτέρω. Καθυστερήσω, μια και έχουμε μόνο μία ώρα στη θέση μας, δίνω το λόγο στους δύο εισηγητές με τέσσερα λεπτά έκαστος θα μας παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Κύριε Χόικμαρκ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους Κιώδης. Δύο συνεδριάσεις έχουν ήδη γίνει. Με τους Κιώδης, τους οποίους και ευχαριστώ. Και αυτό που βλέπω εγώ ως έκβαση είναι να ενσωματώσουμε τα θέματα αυτά τη στείλα στην ε, ε οδηγία για την ανάκαμψη και Εξυγένση, DBRD, BRRD και να τονίσουμε το πώς αντιμετωπίσουμε την τοχευτική ιεραρχία και πώς ε, ερμηνεύουμε το 72B τη CRR, του καρονισμού για, την, για τις κεφαλαίκες απαιτήσει. Υπάρχουν πολλά σημεία συνάντησης, εκ των οποίων ορισμένα έχουν μεγάλη σημασία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλά. Και επίσης συζητήσεις σε σχέση με την μετάβαση από το ήδη υφιστάμενο πτωχευτικό δίκαιο στα θέματα της πτωχευτικής ιεραρχίας ώστε οποιοδήποτε παραλαμβάνει κάποιες ε, ε, πρωτοβουλίες σήμερα να αισθάνεται και για το μέλλον ασφαλής. Για το ΤΙΛΑΚ. Έχουμε ειδικό, ειδική, ειδικό χρέος ε, το οποίο μπορεί να είναι διασωθε, με ίδια μέσα. Αλλά δεν θα πρέπει, από την εμπειρία που έχουμε και από την BRRD, ε, να το πράξουμε αυτό με την, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι ειδικά επιλέξιμο το κεφάλαιο αυτό της διάσωσης με ίδια μέσα. Ότι πρέπει να προτιμηθεί. Πρέπει δηλαδή να διευκρινίσουμε ότι κάθε χρέος είναι διασωτέο με ίδια μέσα, γιατί αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της BRD, ότι δηλαδή δημιουργούμε αυτή την ε, επίγνωση ότι όταν κανείς επενδύει σε μια τράπεζα έχει τους τις ίδιες προϋποθέσεις με τον να επενδύει σε μια οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Πρέπει να διευκρινιστεί λοιπόν αυτό και ταυτόχρονα πρέπει να καθοδηγήσουμε την διαδικασία με βάση και το TILAC το οποίο θα αποτελέσει την ε, βασική αρχή για το MRL. Τις ελάχιστες απαιτήσει δηλαδή ιδιωτικών κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων. Θα έχουμε το TILAC, θα έχουμε το MRL με μια κάποια διαφοροποίηση κάπως. Και είναι ακόμη πιο σημαντικό για ένα λόγο που αντιμετωπίσαμε στην ακρόαση ότι δηλαδή είναι άλλε οι αρχέ. Οι εποπτικέ αρχέ έχουν διαφορετικέ κεφαλαϊκέ απαιτήσει. Οι αρχέ εκαθάρισης άλλε απαιτήσει και MRL, με βάση την MRL. Και άρα ε, τράπεζες οι οποίες έχουν πολύ υψηλό επίπεδο ιδίων κεφαλαίων κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση γιατί τους επιβάλλεται υψηλότερο επίπεδο MRL. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει υψηλό επίπεδο ιδίων κεφαλαίων. Άρα αντίφαση σε σχέση με αυτό το οποίο επιδιώκουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί μια τάξη όπου οι τράπεζε θα μπορούν το MRL να το καλύπτουν με υψηλό επίπεδο ιδίων κεφαλαίων. Είναι βέβαια πολύ λεπτό το ζήτημα. Όπω είπα, είναι διαφορετικέ οι εποπτικέ αρχέ ε, και διαφορετικέ οι προοπτικέ του. Και τώρα έχω φτάσει στα 4 λεπτά και 23 Δευτέρα Πρόεδρε, που δεν ήταν βέβαια αρκετά. Ο Πρόεδρος. Μόνο μία ώρα έχουμε, δεν έχουμε πολλή ώρα στη διάθεσή μας. Μπορούμε όμως να επανέλθουμε. Ο εισηγητής Ιαράρ cr ο Πέτρος Ζήμων, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, στην τοποθέτησή μου σήμερα στην ακρόαση που κάναμε την προηγούμενη φορά, γιατί είναι θέματα τα οποία έχουν και ε, ε, δυναμικό εκρηκτικό, θα έλεγα, και μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Ένα-δύο ζητήματα τα οποία βεβαίως μπορούμε, με τα οποία μπορούμε βεβαίω να αντιπαρατηθούμε, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε για να καταλήξουμε σε μια θέση. Αναλογικότητα λοιπόν. Ήταν ενδιαφέρον για μένα το ότι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή αλλά και ο SSM υποστήριξαν την έννοια της αναλογικότητας ταυτόχρονα όμως επισημένοντας ότι δεν θα την εισήγαγαν στην ε, συχνότητα των κοινοποιήσεων αλλά στο περιεχόμενο για τη συχνότητα των κοινοποιήσεων θα μπορούσε να περιορίσει την ποιότητα της εποπτείας. Και άρα πρέπει να κοιτάξουμε τι συγκεκριμένο περιεχόμενο διευκόλυνση ως προς το περιεχόμενο στις κοινοποίησεις στο πλαίσιο της αναλογικότητας θα πρέπει να εξασφαλίσουμε εφόσον δεν εξαρτηθεί αυτή η διευκόλυνση από την συχνότητα των κοινοποίησεων αλλά από το περιεχόμενο. Και πρέπει εδώ να επισημάνω ότι σε κάθε περίπτωση και συζήτηση που έχω κάνει με όλους τους εκπροσώπους ε, φορέων, ανεξαρτήτως ε, του τι ε, υπόθηκε σε σχέση με τα προβλήματα σχετικά με την πληροφορική. Δηλαδή όταν πια είχαμε αντιμετωπίσει το θέμα της πληροφορικής και δεν ετίθετο πλέον ζήτημα τεχνικών δυσκολιών, όλοι στο ίδιο συμπέρασμα ε, κατέληγαν και επεσήμεναν αυτό το ζήτημα. Ε, απόλυτα κατόφλια σε σχέση ε, με, την αναλογικότητα για τις μικρότερες δηλαδή τα μικρότερα ιδρύματα που θα πρέπει να ευνοηθούν ή με ένα αναλογικό παράγοντα, ένα σχετικό παράγοντα καλύτερα τον οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στην αναλογικότητα. Γιατί, Γιατί ε, μπορεί να έχουμε σε μια χώρα με την κατάταξη αυτή της Επιτροπής ένα ίδρυμα το οποίο θα χαρακτηρίζεται πολύ μικρό ενώ σε μια άλλη χώρα να θεωρείται μέτρο ή και, μεγαλύτερη, και, και μεγαλύτερο και να έχει και συστημική σημασία. Άρα λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να συνδυάσουμε μια προσέγγιση απόλυτων αξιών, με ένα πραγματικό κατόφλι δηλαδή, και μία σχετικής αξίας, αξιολόγηση, η οποία θα σταθμίζει μικρές μεγάλες ε, χώρες και τα ιδρύματα μέσα ανάλογα με το επίπεδο στην κάθε χώρα. Ναι. Επίσης πρέπει να μεριμνήσουμε να μην γίνονται οι δηλώσεις αυτές των δεδομένων επανειλημμένως. Και μάλιστα ε, μάνθηκε το ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών από έναν συνάδελφο εδώ. Θα πρέπει να κοιτάξουμε αυτό το ζήτημα. Επίσης ε, για την Ελβετία και τα τσίζιψη των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχουν ε, διαφορετικά επίπεδα, κατόφλια, από ό,τι μας επισημάνθηκε σε σχέση με αυτά τα οποία είναι προς συζήτηση στις, ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάνουμε μια προσαρμογή όμως στα Τσίζιπς θα πρέπει να αλλάξουμε τελείως συζήτηση σχέση με τη Βασιλεία διότι θα έχουμε διαφορετικό επίπεδο μόχλευσης και για την Ευρώπη αλλά και για την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες σχέση με τα Τσίζιπς. Άρα μάλλον θα πρέπει να αφήσουμε αυτές τις κατά μέρος για, το, για τις προϋποθέσεις του δεύτερου πυλώνα και θα ολοκληρώσω εδώ. Η πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται σε ειδικού ως προς το ιδρύματα κινδύνους που εντοπίζουν οι εποπτικές αρχές Και εδώ η Σουηδία, επισημένω στην ακρόταση, είχε πει ότι συστημικούς κινδύνους μέχρι τώρα στη διαδικασία της ε, εποπτείας τους είχε αφήσει να αλλά βέβαια ε, όταν έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πιστοτικών ιδρυμάτων, τότε μπορούμε να δούμε την κατάσταση διαφορετικά. Άρα αυτοί οι παράγοντες μπορούν να περιοριστούν ε, με την εποπτεία. Αλλά πρέπει να δούμε αν αυτό φέρνει κάποιο αποτέλεσμα επιθυμητό ή όχι. Ευχαριστώ. Και τώρα, πρώτος ομιλητής για το ΕΛΚ. Για δύο λεπτά. Εδώ θα μοιραστούμε τα τέσσερα λεπτά. Ο κ. Μπάλς πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Πολύ ευχαριστώ να λάβω το λόγο για δύο λεπτά τώρα ξεκινώντας γιατί με παρακάλεσε ο κύριος Κάρας να σας ε, μεταφέρω μια σύντομη δήλωση εκ μέρους του. Ε, χρειάστηκε σήμερα να γυρίσει στη Βιέννη σε μια δέσμευση που είχε αναλάβει και δεν μπορούσε να αναβάλει. Ε, ο Ότμαρ Κάρα θεωρεί ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό στάδιο στην εξέλιξη για τα ζητήματα της πιστοτικής ιεραρχίας. Ένα ζήτημα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να σταθμιστούν οι διαφορετικές θέσεις ώστε να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική, σε μια πρακτική λύση. Ο κύριος Κάρας ε, ενθαρρύνεται από την εντύπωση ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση των, του ρόλου των εποπτικών αρχών στην ανταλλαγή δεδομένων και στην άσκηση των ε, δικαιωμάτων τους. Δεν χρειάζεται να γίνεται η δήλωση των ίδιων δεδομένων σε δύο διαφορετικές υπηρεσίες ή αρχές ενώ μπορούν μεταξύ τους αυτές να τα ανταλλάσσουν. Πρέπει να αποφευχθεί η επιπλέον επιβάρυνση από την ε, πολλαπλή δήλωση. Ε, πλατφόρμες με υποστήριξη πληροφορικής ε, πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να είναι σαφείς και οι δομές μεταξύ των αρχών. Στην αναλογικότητα πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία ώστε να μην ε, χρειαστεί να μην κινδυνέψουμε από υπερβολική απορρίθμιση ή από ενίσχυση του κινδύνου και θεωρεί ο κύριος Κάρας ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της συχνότητας των δηλώσεων για τα μικρότερα ιδρύματα. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια διευκόρυνση γιατί πολλές φορές ε, αυτό, ε, αυτή η μεγαλύτερη επιβάρυνση σημαίνει σημαντικές δυσκολίες. οι εξελίξεις με βάση τη Βασιλεία βεβαίως θα πρέπει να αξιολογηθούν και οι δύο fast tracks της ε, ε, CAA ε, θεωρούνται από τον κύριο Κάρας πολύ σημαντικοί παράγοντες για να αποφευχθεί η αποσταθεροποίηση, να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στους διαφορούς παράγοντες της αγοράς που θα τους καθισχάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλετε το να μιλήσετε το δεύτερο μέρος ή μετά. Για ελιστές. Πέντρο Σίλβα Περέιρα για ένα τετράλεπτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω υπενθυμίζοντας την ακρόαση της περσμένης εβδομάδας. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συναγάγει κάποια αρχικά συμπεράσματα. Μπορούμε να πούμε ότι η ευρεία πλειοψηφία απόψεων υποστήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ανανομηνήσεως της ιεραρχήσεως των πιστωτών, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία ε, των ε, χρεών, των παλαιών με κάποιους ε, ενδιαφερομένους που ζητούν μια γρήγορη υιοθέτηση αυτού του τμήματος του νομοθετικού πακέτου. Και είναι κατανοητό αυτό. Πρέπει να δώσουμε σαφήνεια, προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου πάνω απ' όλα στην αγορά. Οι τράπεζες πρέπει να γνωρίζουν ταχύτερο δυνατόν που βρίσκονται τα προβλήματα στον φωτοτήλα και τα MRL και τι ευθύνες και αξιώσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Ακούσαμε και τους ρυθμιστικού φωλεί. Είπαν ότι η νέα κατηγορία χρέους δεν υπονομεύει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλες οι ευθύνε μπορούν να διασωθούν, όλα τα χρέη μπορούν να διασωθούν διεδίων μέσων και δεν θέλουμε να περιορίσουμε το, ε, την αποτελεσματικότητα του εργαλείου διάσωσης με τα μέσα που είναι κάτι που θα καθησυχάζει τα μέλη της Επιτροπής. Όπως συμφωνήσαμε, οι συντονιστές πρέπει να επανεξετάσουν το ζήτημα και να δώσουν το πράσινο φως σε μια διαδικασία ταχείας εγκρίσεως και όσον αφορά την εναρμόνιση της εράρχησης των πιστωτών, κάτι που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο, από ό,τι φαίνεται. Ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ επίγον θέμα που πρέπει να αποφασιστεί. Δεύτερον, όπως είπε ήδη ο Πίτερ Σίμον, θέλω και εγώ να υπογραμμίσω ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην ακρόαση και από πλευράς ρυθμιστικών αρχών και από πλευράς των άλλων διαφορεμένων φορέων συμφώνησαν επί της σημασία της αναλογικότητας Πράγματι πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο να εισέλθει πολύ μεγαλύτερη αναλογικότητα ε, σε αυτό το πακέτο. Όμως πρέπει να πω ξεκάθαρα ότι η αναλογικότητα δεν αφορά μόνο τη διευκόλυνση συλλογής στοιχείων και την αποκάλυψη και διάθεση πληροφοριών, δεν αφορά συχνότητα αποκλειστικά και τη λεπτομέρεια των στοιχείων που δίδονται, όλα αυτά είναι σημαντικά αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά για να πετύχουμε πραγματικά ένα αναλογικό καθεστώς, κυρίως σχετικά με το όλο πλαίσιο διάσωσης. Από τη μία πλευρά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαφέρουν πολύ σε μεγέθη, άρα θα ήταν παράλογο όλες οι τράπεζες ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτών και το συστημικό τους αντίκτυπο να κατηγοριοποιηθούν ε, στο παρομοίω όσον αφορά τι απαιτήσει MRL και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαφέρουν πολύ από τη φύση τους και δρούν στην αγορά ανάλογα με διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα. Όσον αφορά την αλογικότητα, πιστεύω ότι πρέπει να θέσουμε μια σταδιακά αυξανόμενη προσέγγιση όσον αφορά τα MRL, χωρίς υπονομεύουμε την αρχή της διάσωσης μίδια μέσα, του bail Υπάρχουν και προβλήματα ιστορικής φύσεως στον τραπεζικό τομέα και κάποιες τράπεζες έπρεπε να αντιμετωπίσουν νέες απαιτήσει πολύ πιο αυστηρές που επευλήθησαν τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν θεσπίζουμε ένα νέο επίπεδο απαιτήσεων. Κλείνοντας θα πω ότι το θέμα των MPLs των κόκκινων δανείων σχετίζονται ε, με αυτό το πακέτο και πρέπει να εξεταστούν. Αυτό αναφέρθηκε εδώ στην ακρόση και πρέπει να το επανεξετάσουμε διότι είναι υψής της σημασίας. Άμα μάλιστα συγκρίνουμε αυτό το θέμα και με τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Ο κ. Φόξ για το ECR έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ECR ορίζει την ενσωμάτωση των διεθνών προδιαγραφών στο CRR2 και το CRD5 και συμφωνούμε με τα περισσότερα από τα προτινόμενα. Με τα χαράς βλέπουμε ότι το FRS 9 προωθείται τετάχιστα και χθε έγινε η πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών επ' αυτού. Όμως πρέπει να αποφασίσουμε ποια μεταβατική προσέγγιση θα ακολουθηθεί και παροτρύνω να διεξαχθεί ανοιχτή και διαφανή συζήτηση, τους ώστε να καταλήξουμε στα καλύτερα δυνατά συμπεράσματα, αντί να διαλέξουμε την απλούστερη λύση, κάτι που προτείνεται από την, από την EBA, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, στη συνεδρίαση. Όποια λύση και να βρούμε, θα πρέπει να την λάβουμε υπόψη αυτή τη λύση, κάνοντας αξιολόγηση συνεπειών. Ήταν καλή συζήτηση που έγινε στην ακρόαση της πέρασμενης εβδομάδας. Είναι σαφές ότι υπάρχουν ακόμα κάποια περίπλοκα ζητήματα προς συζήτηση. Επί παραδείγματι, οι τα περισσότερα κατώμενα ομόλογα δεν θεωρούνται σαν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ε, υπό την ερμηνεία την παρούσα του CRR. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είπε όμως ότι θα γίνει επέκταση του πεδίου αναγνωρίζοντας και το ότι δεν ταιριάζει η λήξη αυτών των ομολόγων για την γίνεται σωστή κάλυψη. Αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση. Ε, πρέπει να δούμε τη σφαιρικότερη εικόνα. Ε, να σημειώσουμε ότι πολλά θέματα δεν συζητήθηκαν και δεν ακούστηκαν στην προηγούμενη ακρόαση. Παραδείγματο χάρη, μάθαμε ότι 13 κράτη-μέλη ζήτησαν διαγραφή των προτινόμων τροπολογιών των άρθρων 7 και περί εξαιρέσεων από ρευστότητα και κεφαλουχικές απαιτήσει για το CRR. Ε, αυτό γιατί συζητήθηκε. Πρόεδρε, ο συνάδελφο Ζαϊκ Καμάλ δυστυχώ δεν μπορεί να παραστεί σήμερα η συζήτηση, όμω θα στείλει τα δικά του σχόλια όσον το, πακέτο, το τμήμα BRD του πακέτου στον εισηγητή. Thank ε, ε, Εμείς ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε και βγες παρατηρήσει εκ μέρους της συναδέλφου Σιλβί Γκουλάρ να σας πω επιλέξει τι έχει να πει. Ότι ήρθε η ώρα να λάβουμε υπόψη το ότι η Τραπεζική Ένωση είναι μία αρχή. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι είδου επιλογές μπορούμε να έχουμε για περιχαράκωση, ιδίω όσον αφορά το εσωτερικό MRL. Οπότε σε μερικές περιπτώσεις θα πρέπει να κάνουμε κάποια ανάλυση όπως το NDA και αυτό το μορατόριο που υπάρχει όσον αφορά την, ε, το άρθρο 55, επίλυση των διαφορών. Το άρθρο 55 λοιπόν για συμβατικές σχέσεις με τρίτες χώρες. Οπότε ίσως θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι επαφέ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι χρήσιμε όσον αφορά το calibration και τις σχετικές απαιτήσεις για τη μέτρηση και το πώς θα βρούμε την ισορροπία μεταξύ προβλεψιμότητας και σταθερότητας για το πώς θα έχουμε επίσης ρευστότητα και χρηματοδότηση της οικονομίας. Το θέμα είναι το πώς θα μπορούμε να δούμε τις δυνατότητες της να ανταγωνιστούν με θεμητούς όρους εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, αυτό τώρα μου δίνει την ε, σκητάλη για να σας πω εγώ ότι πρεσβεύω για το CRR και το CRD, τον κανονισμό και την οδηγία, είτε εδώ πέρα τι θέλει το ρήτημα όσον αφορά το πώς θα μεταχειριστούμε το software, αυτό το λογισμικό. Ρώτησα και δεν έλαβα απάντηση που με καλύπτει, γιατί προβληματιζόμαστε μια που στο δίκαιό μας το λογισμικό θα πρέπει από το πρώτο tier, το πρώτο, το πρώτο επίπεδο του, του κεφαλαίου να εκπέσει. Και είναι θέμα τώρα τι θα γίνει σε περίπτωση πτώχευση, αν θα πρέπει να υπάρξει διαφορεμένη μεταρρύθμιση. Άρα, να, το πρώτο γιατί δεν μπορεί αυτό να γίνει μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι το εξή, ότι Φερρυπίν στη ΣΥΠΑ το software δεν χρειάζεται να εκπέσει ή να αφαιρεθεί. Άρα αυτό είναι μειονέκτημα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Καλά, λέμε ότι στην Ευρώπη εμεί σκεφτόμαστε διαφορετικά. όμω αναδύεται άλλο πρόβλημα. Δηλαδή ότι, ότι έχουμε αυτό το καθεστώς τη ισοτιμίας, ισοδυναμίας, αντιστοίχηση ε, για, για, τη, σημασία του θέματος αυτού. Οπότε έχουμε τις αμερικάνικέ τράπεζε που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επενδύουν στο λογισμικό πολύ περισσότερο από όσο οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Άρα νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το μελετήσουμε ή να αλλάξουμε το καθεστώς της ισοτιμίας ή θα πρέπει να γίνει με μεταβολή του καθεστώς και για τις ευρωπαϊκές τράπεζες γιατί είμαι πεπισμένη ότι με όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στα τραπεζικά όσον αφορά τα fintech ε, θα πρέπει κανείς να είναι μέσα στις εξελίξεις. Τώρα δεν είμαστε. Δεν νομίζω ότι μπορούν τα χρηματοδοτικά ιδρύματα να το κάνουν αυτό. Ε, ε, οι τράπεζες όπως οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που να ανταγωνιστούν για το fast tracking συμφωνώ με τόσο που ο κύριος Ζήμων ότι δηλαδή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει κάποιο είδους ομαλή μετάβαση χωρίς κάποιο είδους αθέλητες ε, συνέπειες λοιπόν αυτό να γίνει εφικτό αλλά να προσέξουμε για το τι θα γίνει πώς θα είναι αυτή η μεταβατική περίοδος. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι κάτι όλος νέο. Θα πρέπει να δούμε αν θα συντρέχει εδώ αναλογικότητα, να κάνουμε τις μελέτες επιπτώσεων, οι οποίες ε, είναι αρκετά συγκεκριμένες. Είναι θέμα μέσων όρων. Και επαναλαμβάνω, αν κανείς έχει τα πόδια στο ψυγείο και το κεφάλι στο φούρνο, καλή είναι η μέση θερμοκρασία. Αλλά κάποιος συνεχίζει να μην αισθάνεται τόσο άνετα. Οπότε για να δούμε τι λένε οι μελέτες όσον αφορά τη σύγκριση των επιχειρηματικών μοντέλων μεταξύ μικρών, μεγάλων ε, τραπεζών και να βγει μια ε, λογική ε, σύγκριση. Απ, τέλειωσε ο χρόνος μου όμως. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και δίνει το λόγο στον κύριο Ντεμάζη για δύο λεπτά για την ΚΟΕ. Uh, yeah, Καλημέρα. Ωραία, πολύ καλό είναι αυτό το ότι μοιράζεται ο χρόνο αγορεύσης. Όσον αφορά την ε, διακριτική ευχέρεια της εποπτείας, συμφωνούμε όσον αφορά το κεφάλαιο και θα πρέπει οι υποπτικές αρχές να έχουν την αρμοδιότητα να επιβάλλουν κάποιο είδους υποχρεωτικές ε, ε, απαιτήσει και όχι μόνο κατευθυντήριε. Να μπορούν επίση να έχουν τέτοιου είδους μακροπροληπτική εποπτεία Ακριβώ όπω τα είπαμε για την περασμένη εβδομάδα στην ακρόαση. Τώρα όσον αφορά την ιεράρχηση των ε, ε, πιστωτών θα πρέπει να δούμε το τι μέσα θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρεωστικά μέσα τα οποία ξεκινούν από το κάποιου κανόνε γιατί κάποια προϊόντα στην πράξη δεν μπορούν να περάσουν μπέιλιν διάσωση Οπότε το fast tracking για αυτά δεν νομίζω ότι προς το παρόν γίνεται. Όσον αφορά τα μέσα, τα χρεωστικά για τρίτες χώρες, θα πρέπει να τύχουν άλλε μεταχείρισεις και αν θέλουμε να έχουμε εξαιρέσεις, να δούμε το ότι μπορεί αν υπάρχει κάποια διαφορά να επιληθεί με κάποιο είδους άνω όρια. Τώρα όσον αφορά την προληπτική εποπτεία και τη σχετική ε, ρήτρα ε, να γίνει αυτή τη ρήτρα η αξιολόγηση, αλλά διαπιστώνουμε ότι σε περιπτώσεις που στριμώνεται μια τράπεζα, ένα οργανισμός, τότε ο ιδιωτικό τομέας δεν μπορεί πάντοτε να πετύχει αξιόλογες επιδόσεις. Υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στον ε, κλάδο, οπότε αυτή η ρήτρα ανακεφαλαιοποίηση νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά στο παρελθόν Άρα εδώ θα πρέπει να το ξανακομεντιάσουμε προσεκτικά και για το MRL είπαμε ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το TLAC, με τι κάτι ισχύει, να επιληθούν τα προβλήματα και οι αρχές επίλυσης διαφορών επίσης να προσέχουν και να εφαρμόσουν κάποια διαρθρωτικά μέσα, εάν χρειάζεται. Ο κύριος Μακάρτη. Ευχαριστώ, όπως είπα και στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το τραπεζικό πακέτο. Καταρχήν είμαστε υπέρ οποιασδήποτε προσπάθειας περιορισμού του κινδύνου και να μην κοινωνικοποιούνται οι ζημίες. Έχουμε την πρόταση της Κομισιόν για την οδηγία και τον κανονισμό πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Όμως έχουμε εδώ πολλά παραθυράκια, πολλές αποκλήσεις από τα διεθνή πρότυπα. Άρα θα πρέπει να κλείσουμε τα παραθυράκια και αυτού του είδους οι αποκλήσεις να διορθωθούν. και να δούμε τι θα γίνει με την, ε, με την μόχλευση, το ποσοστό αυτής ε, μας προβληματίζει και θεωρώ ότι το 3% είναι πολύ χαμηλό και ε, πολλοί γνωμολόγοι λένε ότι κάνει, χρειάζεται πολύ, κάτι πολύ παραπάνω για τις τράπεζες όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών ούτω ώστε να, η, η μέτρηση να έχει λιγότερο ποσοστό λάθος. Άρα θέλουμε να το χρησιμοποιήσουν και οι ρυθμιστικές αρχές και οι τράπεζες. Για το τίλακ τώρα γενικά θέλουμε να αυξηθούν οι κεφαλικές απαιτήσεις για τις συστημικές τράπεζες, να μην έχουμε περίπλοκες έννοιες όπως το τίλακ Δεν αποδίδουν όταν ε, η κρίση χτυπήσει την πόρτα. Και όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο και την περιουσία της τράπεζας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί το ότι θα έχουμε τα σωστά κριτήρια επιλεξιμότητος. Και θα πρέπει να δούμε τι κατησχύει το τι ή άλλο πρότυπο όταν έρθει η κρίση και να υπάρχουν αυτές τις κανθήριες γραμμές για το κεφάλαιο και το IFRS 9 θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη την πρώτη χρονιά και να μην αποκλίνουμε από τα διεθνή πρότυπα, ό,τι και να κάνουν οι Αμερικανοί. Να γίνει προετοιμασία για αυτούς τους κανόνες λογιστικής, τους νέους και από το χρόνο είπαμε θα έχουμε αυτή την μεταβατική περίοδο των πέντε ετών. Πολύ μακρά περίοδος. Να προσέξουμε αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ για τους πράσινους. Ούρτανσον για δύο λεπτά. Και μετά ο Φίλιπ Λάμπερτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα αναφερθώ σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα για την ιεράρχηση της φερικαιότητας και το ε, όλο καθεστώς ε, για τη διάσωση. Για το θέμα της φερικαιότητας βλέπουμε την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να ενισχύσουμε την αρμόνιση της ιεράρχησης των πιστωτών αλλά τρία σημεία της γνωμοδότησης πρέπει να εξεταστούν. Πρώτα απ' όλα η δημιουργία γενικού κανόνου για προτίμηση καταθετών, μετά διάταξη που θα λέω ότι όταν υπάρχουν μέσα χρέωσης που θα πρέπει ε, εκπνέουν, θα πρέπει να οι νέε εκδόσεις ομολόγων πρέπει να ευθυγραμμίζονται σωστά όπου εδείκνεται με το καθεστώς που προβλέπεται για τη νέα τάξη ε, νέων ε, μέσων για την αρμόνιση των διαφόρων μέσων και την αξιολόγηση των, των στοιχείων παθητικού, αυτά θα πρέπει να συζητηθούν. Μετά, όσον αφορά το καθεστώς διάσωσης, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα πιο αξιόπιστο καθεστώς και γι' αυτό είναι σημαντικό υπολογίζοντας ε, των στοιχείων παθητικού και διάσωση ίδια μέσα να βάλουμε το 8% για να υπάρχει πρόσβαση στο Ταμείο Διάσωση. Αλλιώ δεν θα είναι αξιόπιστο το καθεστώ. Και ανησυχούμε κατά πόσο ο υπολογισμό των στοιχείων ενεργητικού και του ποσοστού μόχλευση μα φτάνει στο 8%. Και όπως είπε και το Συμβούλιο περί διασώσεως πρέπει να έχουμε 8% ε, ποσοστό στοιχείων παθητικού και άλλα δύο να πούμε ότι ε, Ανησυχούμε για το θέμα των προσανατολισμών του πυλώνα 2. Πρέπει να ενισχύσουμε τις εξουσίες του εποπτικού φορέα με καλύτερο αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Όταν δεν υπάρχει συμμόφωση με κατευθυντήρια γραμμή, πρέπει αυτή να μεταμορφώνεται σε απέτηση. Ο συγκεκριμένο χρονισμό τη διαδικασία είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί, είναι σημαντικό. Τέλο, και θα κλείσω γιατί δεν έχω χρόνο, για το νέο εργαλείο παγώματο, το moratorium, θα πρέπει να δούμε μήπως μπορούμε να έχουμε εξαιρέσει για κάποια στοιχεία παθητικού, κυρίως για τις νομικές επιχειρήσεις, για να μην ε, τους περιορίζουμε στις αστηριότητες. Αυτά είναι κάποια σημεία τα οποία ήθελα να θέσω. Φίλιπ Λάμπερτς. Καλημέρα. Θα ήθελα να είναι ένα πακέτο μείωση των κινδύνων. Είναι. Το θέμα είναι για ποιον όμως. Ε? Η μείωση του κινδύνου αφορά τους μετόχους και τους διαχειριστικούς φορείς των τραπεζών ή για τους φορολογούμενους. Και αυτό είναι κάπως ασαφές για μένα. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να δείχνουν ότι είναι ένα πακέτο μείωση του κινδύνου περισσότερο για τους μετόχους. Δύο παραδείγματα. Ένα το έθεσε ο Φάμπιο πριν. Όταν δεσμεύεις ουσιαστικά και περιορίζεις το ρυθμιστικό φορέα και τις υποχρεωτικές απαιτήσεις μεταμορφώνεις σε προσανατολισμούς, τότε αυτό μειώνει το κίνδυνο για τους μετόχους. Αλλά αυξάνεται ο κίνδυνο για τους φορολογούμενους. Παρομοίως. Το ποσοστό μόχλευσης ήταν μια απλή έννοια. Τώρα μιλάμε για έκθεση, για μέτρο έκθεση σε μόχλευση. Και αυτό μου μυρίζει σαν ε, στοιχεία ενεργητικού με στάθμιση για το κίνδυνο. Ε, Μπορεί να το χρησιμοποιήσουν ε, αν θέλουν οι τράπεζε τελικά, υπερβολικά. Εγώ είμαι ένα απλό άνθρωπο. Όταν χρηματοδοτείς μια επιχείρηση λοιπόν, μέσω του ενός, ε, με 3% με κεφάλαιο και 97% με χρέος, που να προσπαθήσει να το στρίψει από εδώ, από εκεί, αλλά τελικά ε, το βρίσκω πάρα πολύ εύθραυστο σαν προσέγγιση. Άρα θα πρέπει να έχουμε το θάρρος και να πούμε καλώς ας επιβάλλουμε αυστηρότερες προδιαγραφές για τη μόχλευση θα χρησιμοποιήσουμε τα προτινόμενα μέτρα βέβαια, αλλά όσον αφορά την επιβολή πραγματικών απαιτήσεων κεφαλουχικών θα πρέπει να είμαστε αυστηρότεροι. Κάποιο είπε ομά. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να είμαστε ασφαλείς παρά να διακινδυνεύουμε και να το μετανιώνουμε μετά. Το λέω σαν φορολογούμενος. Λοιπόν, αν θέλουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο, δεν, θέλουμε, δεν βλέπω να μειώνεται για φορολογούμενους. Δεν, η πειθαρχία της αγοράς δεν πληρώνεται από τους ε, ε, φορολογούμενους. Αν κάποιος κάνει ανοησίες πρέπει να τιμωρείται με τα δικά του χρήματα. Αυτή είναι η οικονομία της αγοράς. Μ' αρέσει να ζω στην οικονομία της αγοράς, αλλά με θλίψη λέω ότι πολλά από αυτά που βλέπω στο πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατευθύνονται περισσότερο προς παλιές καλές ή μάλλον κακές ημέρες που προηγήθηκαν της κρίσης. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να αντέξω στον, στον πειρασμό να σας πω ότι αυτό διακρίνει μια τράπεζα από την υπεραγορά δεν είναι μόνο ότι έχουμε τη διαχείριση και τους φορολογούμενους, τις χειριστικές αρχές, αλλά έχουμε και τους καταθέτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καταθέτουν τα χρήματά τους για να πληρώσουν μισθούς. Οι μικροεπενδυτές. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία που περιπλέκει περισσότερο την κατάσταση. Εγώ τους αποκαλώ πελάτες πελάτες είναι και πρέπει να αποφασίζουν με ποιον ε, συναλλάσσονται. Είναι δική τους ευθύνη επίσης. Υπάρχουν καλές επιχειρήσεις και κακές επιχειρήσεις και θα πρέπει κανείς να μπορεί να διαλέξει. Δεν αγοράζω από οποιονδήποτε. Δεν θα εάν θα πρέπει να υπόκειται ο πελάτης της αγοράς ε, σε πειθαρχία της αγοράς, δεν θα έχουμε την προστασία του καταθέτου. Θέλετε να μπούμε σε συζήτηση, υποστηρίζω την προστασία των καταθέσεων μέχρι κάποιο βαθμό, όχι απεριόριστα. Καλώς, έξοχα. Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι εισηγητής Σκιώδης και για τα δύο ζητήματα και θα μακρηγορήσω κάπως. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι το πρώτο δεν είχα τη δυνατότητα να ακούσω στην ακρόαση κάποιο νομικό εμπειρογνώμονα για να δω ποιες θα μπορούσαν συνέπειες σε κάποια κράτη-μέλη, συνέπειες σχετικά με την σωμάτωση του BRD και το σύστημα ε, σε, σε περίπτωση διάσωσης τραπεζών. Σε κάποιες χώρες συνταγματικώς προβλέπεται το δικαίωμα προστασίας των αποταμιεύσεων. Θα ήθελα λοιπόν να έχω την άποψη της νομικής άποψης κάποιων ε, εμπειρογνωμόνων για να δούμε ποια θα είναι τα προβλήματα εκεί που έχει εφαρμοστεί ήδη το Μπέιλιν στη διάσωση διότι δεν εφαρμόστηκαν παρομοίως στις ίδιες χώρες τα μέτρα. Στην Ιταλία που χρησιμοποιήθηκε αυτό το μέτρο δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Αυτό είναι το σημείο. Ε, λοιπόν, αυτό επιφέρει περισσότερη αστάθεια, διότι καλούνται πάντα οι φορολογούμενοι να πληρώσουν οι συνεισφέροντες και οι αποταμιευτές πολύ συχνά εν άγνοιά τους μπαίνουν σε καθεστώς που τους τιμωρεί. Δημιουργείται αβεβαιότητα για τις τράπεζες και έτσι μετά οι αποταμιευτές δεν καταθέτουν ε, ε, να τα πηγαίνουν, πηγαίνουν τις καταθέσεις τους είτε σε μεγαλύτερες τράπεζες είτε σε άλλες χώρες. Ε, βλέπουμε αν δείτε τι γίνεται τις ροές των καταθέσεων και των κεφαλαίων. Και αυτό είναι κάτι αξιόμεμπτο σαν κατάσταση. Όσον αφορά το συγκεκριμένο, ζητήσαμε διαφάνεια όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τα MRL και σε περίπτωση διάσωσης πιστεύουμε ότι οι αρχές μαζί με την Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει ανάλογα με τις ανάγκες εμπιστευτικότητας για ασφάλεια των αγορών να κινούνται. Σύμφωνα με όταν όμως δεν είναι πλέον ε, ευαίσθητες πληροφορίες να δημοσιεύονται σε αποφάσεις. για όσον αφορά τη διάσταση των τραπεζών. Υπάρχει διαφάνεια. Στην κατηγορία του senior debt είδα το θέμα αυτό. Βλέπ, συναντήθηκαν διάφορους stakeholders για να το συζητήσω μαζί τους. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε περίπτωση όπου αυτά τα νέα προϊόντα διατεθούν σε συνταξιωτικά ταμεία, σε ασφαλιστικά ταμεία, αποσφαλιστικά ταμεία Ίσως να δημιουργείται ένα θα έπρεπε να είναι πιο συντηρητικέ επενδύσει. Ένα κομμάτι των επενδύσεων να είναι πιο συντηρητικό. Αντί να μπαίνουν τα χρήματα ε, σε επενδύσει που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διαδιάσωση. Οπότε δημιουργούνται συστημικά προβλήματα διαχείριση. Τώρα, όσον αφορά τι απαιτήσει κεφαλουκικέ, πιστεύουμε ότι η προσέγγιση είναι εσφαλμένη. Διότι το σύστημα επικεντρώνεται υπερβολικά σήμερα επί των δραστηριοτήτων πιστώσεων αντί των assets δευτέρου και τρίτου επίπεδου. Και αυτό δημιουργεί ασφαλμένη εικόνα του τραπεζικού συστήματος σήμερα στην Ευρώπη. Ευνοεί τράπεζες που, είναι πιο, που κάνουν πιο επικίνδυνες επενδύσεις, ενώ οι λιγότερο, οι πιο συντηρητικές βλέπουν να επιδεινώνεται η κατάστασή τους. Άρα θα σκοτώσουμε ένα κομμάτι του τραπεζικού συστήματος έτσι και διευκολύνουμε ένα κομμάτι των τραπεζικών που θα πρέπει να τιμωρηθεί μετά την κρίση. Για μας είναι σημαντικό αυτό. Πέντε δευτερόλεπτα. Να αποφύγουμε τι, όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα, να υπάρξει εξαίρεση όσον αφορά το κίνδυνο. Θα πρέπει εκεί να έχουμε μια θέση πολύ πιο προσεκτική όσον αφορά αυτών των μέτρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριο Σάνη. Μια σύντομη μεθοδολογική παρατήρηση. Θα πρέπει να παρέμβουμε γιατί το ΕΝΕΦ έχει περισσότερα μέλη. Πρέπει να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι δεν μπορείτε να μας αφήνετε δεύτερους. Κάτι ακόμη τώρα για τις ε, προτάσεις αυτές. Ο Φιλίπ αναφέρθηκε νωρίτερα στους στόχους. Δύο είναι οι κύριοι στόχοι που θα πρέπει να επιδικήσουμε όχι η πρόταση αυτή, τουλάχιστον όπως βλέπω εγώ τα πράγματα. Ο πρώτος είναι να γίνει μια διόρθωση έστω και μερική σε σχέση με σφάλματα προηγούμενα στην σύσταση, στην κατασκευή της Τραπεζικής Ένωσης, εάν βεβαίως ήταν τυχαία και όχι εσκεμμένα τα σφάλματα αυτά. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τα διορθώσουμε τώρα. Και ο δεύτερος, πιο γενικός στόχος, θα πρέπει να είναι αυτό στο περιορισμό του κινδύνου, αλλά εν γέννη περιορισμό του κινδύνου, στον οποίο είναι εκτεθειμένο όλο το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να θεωρηθούν προνομιούχοι μόνο ορισμένοι κάτοχοι χρέους των τραπεζικών ιδρυμάτων ή μόνο κάποια άλλη κατηγορία. Μια καλή συνεργασία, μια καλή δουλειά σημαίνει γενικά μείωση του κινδύνου για όλους τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζονται από την δράση και το τραπεζικό σύστημα εν γέννη. Ε, σε σχέση λοιπόν με τις προτάσεις, όπως είπα να διορθωθούν σφάλματα και στρεβλώσεις της Τραπεζικής Ένωσης και της ε, μέχρι τώρα νομοθεσίας. Είναι ουσιώδου σημασία να θεσπιστεί ένα σύστημα και αναφέρομαι εδώ βέβαια και στην ε, μεταφορά στην Ευρώπη του ΤΙΛΑΚ όσο το δυνατόν πιο ομοιογενές ένα σύστημα το οποίο να επιτρέπει λιγότερη ευχέρεια ακόμα και από τις αρμόδιες αρχές ε, επαγρύπνησης και γιατί, γιατί με την Τραπεζική Ένωση και την ε, ενιαία μοναδική αρχή εποπτείας ε, βιώνουμε αυτή τη στιγμή ορισμένε περιπτώσεις και ιδιαίτερες καταστάσεις οι οποίες ομολογώ πως με προβληματίζουν ως προς την ιδέα της ε, εφαρμογής των ίδιων αρχών επαγρύπνησης για όλα τα ιδρύματα από τη μία αυτή αρχή. Ποιος είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι να προκύψουν στρεβλώσεις. Το ανέφερε ο Φάμπιο Ντεμάζη νωρίτερα. Σε σχέση με την Τίλα και τη Μέρλα. Από την περιπτωσιολογική προσέγγιση. Και τη μεγαλύτερη ευχέρεια που θα έρχει η αρχή επαγρύπνησης με τον κίνδυνο να προκύψουν καταστάσεις που θα έχει επηρεάσει μια πολιτική επιλογή και όχι ο τεχνικός χαρακτήρας της κατάστασης και της ανάγκης για προστασία των συμφερόντων των πολιτών ή του ε, όποιου έχει επενδύσει στο τραπεζικό σύστημα, αλλά που θα έχουν ακολουθήσει μια πολιτική καθοδήγηση. Και μια τελευταία παρατήρηση για τη δέσμη αυτή, η δημιουργία ενός νέου συστήματος ε, χρέους που έχει να κάνει με τους μη προνομιούχους με εξοφλητική προτεραιότητα, νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη... Ε, ε, έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη αυτή στρεβλωτική δυνατότητα του BRRT, δηλαδή να υπάρχουν συστήματα μέσα καλύτερα, που θα αποτελούν ένα ε, δίκτυ προστασίας, μια ζώνη ανάσχεσης και προστασίας ανάμεσα στα ε, προνομιούχες και μη στους προνομιούχους και μη προνομιούχους χρεωστικούς τίτλους. Προστατεύεται δηλαδή ο επενδυτής σε σχέση με ένα βαρύ σφάλμα της BRRD που ήταν κατά την ε, δική μου θέση η αναδρομικότητα σε σχέση με εκείνους που μπήκαν ε, εκ των υστέρων για να επωφεληθούν από χαμηλέ τιμέ. και άρα τώρα βρισκόνται σε με... καθεστώς μεγαλύτερης προστασίας. Ε, επίσης, όπως είπε και ο Φιλίπ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο του κινδύνου ε, και σε σχέση με, τις, ε, με το δημόσιο χρέος. Υπάρχει ο κίνδυνος μια στρέβλωση ή και πίεσης, στρε δηλαδή μεγαλύτερου για τις ε, τράπεζες σε σχέση με τους ε, επενδυτές αυτού του δημοσίου χρέους. Άρα χρέος, ε, πίεση μεγαλύτερη για το κρατικό χρέος που ήδη βρίσκεται σε συνθήκες δύσκολες αυτή τη στιγμή. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ξέρετε για τη σειρά που αναφέρατε, η ΕΝΕΦ και τα λοιπά. Ακολουθούμε γενικά τη σειρά που έχουν οι πολιτικές ομάδες στην Ολομέλεια. Και έτσι πρέπει να αντικατοπτρίστε και η συμμετοχή του στις κοινοβουλευτικέ επιτροπές, αν και αυτό δεν ισχύει πάντα. Μα ήταν οι ομιλητές σε διαφορετική σειρά. Η ΕΝΦ ήταν πριν από το EFTD, ε στο mail που μας έστειλε η γραμματεία. Μια παρατήρηση έκανε, πας περιπτώσει. Πρόεδρος. Κύριος Μπάλτς, με άλλα δύο λεπτά τώρα. Παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να υποστηρίξω ρητά τον συγκητή μας τον κύριο Χεκμάρκ σε σχέση με την πειθαρχία και την αγορά που επισημαίνει ο Γκούναρτ. Ε, τρεις εκθέσεις περιορισμού του κινδύνου έχουν βασικά το ίδιο χαρακτηριστικό και πρέπει να το υπογραμμίσουμε ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε με κριτικό βλέμμα εάν με το έμρε αρκεί το επίπεδο το οποίο προτείνεται με το ελάχιστο του 8% στο σύνολο των ε, υποχρεώσεων ε, που θα πρέπει να ξανασυστηθεί πιστεύω. Δεύτερον, ο τρόπος υπολογισμού, η διακριτική ευχέρεια καλύτερα από την εποπτική αρχή ε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσουμε σε πέντα χαμηλότερα από το status quo σε σχέση με την TILAC. με τις ρυθμιστικές ε, προδιαγραφές της ΕΜΡΕΛ. Και τρίτον, οι δυνατότητες για παρέκκληση σε σχέση με τη σειρά πάλι δεν θα πρέπει να είναι σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προτείνει η ΤΙΛΑΚ. Για τα ίδια κεφάλαια τώρα. Θα ήθελα να υποστηρίξω τόσο είπε ο Ζημών ε, για την αναλογικότητα. Νομίζω ότι δεν φτάνει μέχρι το βαθμό που θα θέλαμε η πρόταση της Επιτροπής. Θα χρειαζόταν κάποιες ε, τροποποίησεις, όχι μόνο ως προς την διατύπωση της υποχρέωσης κοινοποίησης, αλλά και πέραν αυτού του των προδιαγραφών που θα πρέπει να ισχύουν για όλες τις τράπεζες, για όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, μικρά ή μεγάλα, και όχι μόνο για τα μεγάλα επίσης οι επενδυτικές τράπεζες για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη υποστήριξη στην ανάπτυξη ε, της οικονομίας πρέπει να ανοίξουμε τους οριζοντές μας σε σχέση με τις επενδυτικές τράπεζες. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω, να ενθαρρύνω τον ε, συνάδελφο και εισηγητή Πέτερ Ζήμων για πιο φιλόδοξες απαιτήσει ε, που θα ξεπερνούν το status quo. Για τον κύριο Σίλβα Περέρα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι συντονιστές πρόσφατα συζήτησαν το θέμα του fast tracking για τις τράπεζες και έχουν αποφασίσει με βάση τις αρχές της πλειοψηφίας. Ευχαριστώ. Thank you. I have also request... Ευχαριστώ, λέω. Πρόεδρος ο Μάρκος Φέρμπερ όμως έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, ναι. Να το catch the eye που έχουμε δώσει. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, πρέπει να δούμε καταρχάς αν αξίζει το όνομα αυτό το πακέτο που έχει τον τίτλο περιορισμός του κινδύνου ή αν τελικά δεν συμβάλλει στον περιορισμό του κινδύνου. Και θα υπογραμμίσω με ιδιαίτερη έμφαση τα όσα είπε ο κύριος Χέκμαρκ. Δεύτερη παρατήρηση. Αναλογικότητα. Η Επιτροπή μέχρι τώρα έναν δείκτη μόνο έχει αναφέρει. Τον όγκο του ισολογισμού δηλαδή δεν αρκεί για μένα. Γιατί ο όγκος ε, του ισολογισμού δεν δίνει στοιχεία, ε, ε, ενδείξεις για την έκθεση κίνδυνο μιας τράπεζας. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους λοιπόν αξιολόγησης, διότι όπως είπα ο όγκος αναλόγως του μεγέθους του κράτους μέλους μπορεί να δίνει διαφορετικές και μάλιστα εσφαλμένες <coughs> ενδείξεις για την έκθεση σε κίνδυνο. Άλλα κριτήρια χρειάζονται λοιπόν. Πρέπει να αναπτυχθούν φερπίν, ε, περιφερειακή αρχή, ε, μη υπερσυνοριακές δραστηριότητες, ε, ε, δομή επενδυτών, θεσμικοί επενδυτές ή όχι, Διάφορα κριτήρια λοιπόν που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μέσα σε ένα δελτίο και πολύ ευχαριστώ να συνεργαστώ και εγώ έτσι ώστε να έχουμε ένα όσο το δυνατόν συνεκτικό ε, σύστημα μια πρώτα συνεκτική που να μπορεί να εφαρμοστεί σωστά σε κάθε κράτος μέλος και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορεί να σταθμίσει αυτούς που έχουν χαμηλή, χαμηλό επίπεδο ε, ε, όγκο ισολογισμού ή απλή δομή επενδυτών να μην αντιμετωπίζονται πάντα με τον ε, ίδιο τρόπο, διαφορετικά να αξιολογεί το κίνδυνο του σε πάση περιπτώσει. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο, νομίζω, για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και... Ε, ζητώντα συγγνώμη από την Επιτροπή, θα τη πω ότι αυτό που μα προτείνει δεν μα βοηθάει, δεν βελτιώνει δηλαδή καθόλου την κατάσταση. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να στεί κανεί άλλο το λόγο στη διαδικασία Καριστιάη. Δίνω λοιπόν το λόγο και πάλι στους εισηγητές. Δύο λεπτά έκαστος κύριε Χέκμαρκ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι να, πρόκειται να ζητηθεί σύντομα το fast tracking. Όχι, ούτε εγώ την Πεστρομά έχουμε κάτι να πούμε εναντίον του fast track. Έτσι κι από φιλοσοφικής πλευρας όλοι fast track κινούμεθα. Αλλά αλλά να μην το κάνουμε ε, με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην ξέρουμε τι κάνουμε γιατί υπάρχουν κοινά σημεία σε αυτά τα πακέτα και για να καθορίσουμε την ιεραρχία τη σειρά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα κριτήρια του MRL εκεί σε αυτά τα σημεία του πακέτου το οποία είναι του κ. Ζήμων το 72B ας πούμε και συνάδελφοι όλοι είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και προκαταρκτικές συζητήσεις αλλά επίσης είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί αυτό που θα σας πω για πολλωστή φορά ότι αν δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την BRD θα πρέπει όλα αυτά να είναι τέτοια που να επιδέχονται διάσωση με ίδια μέσα. Θέλουμε να εξαιρέσουμε μεγάλα κομμάτια παθητικού από αυτή την διάσωση. Έτσι όμως υπονομεύουμε την πειθαρχία στην αγορά. Αυτό το οποίο το BRD ε, σκόπευε και αυτό είναι πολύ σημαντική κατάκτηση. Για μένα, επομένω αυτό είναι ε, ρίσκο και συμφωνώ με τους πράσινους. Τέλος πάντων, οι αυτοί συμφωνούν με μένα, δεν έχει σημασία. Αλλά είναι σημαντικό να μείνουμε πιστοί στην πειθαρχία της αγοράς. Εγώ θέλω κάτι τέτοιο να το εξασφαλίσουμε ακόμα και όταν συζητούμε για το fast track και την ιεράρχηση, τη σειρά. Ευχαριστώ. Παρατηρήσεις εκτός μικροφώνου. Θα πρέπει να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε, λέει ο πρόεδρο σούπερ μάρκετ ή τράπεζα. Και τελικά δεν υπάρχει πειθάρχηση στην αγορά. Έτσι, αν δεν ξέρω. Κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Χόκμα, ταυτόχρονα με τον Πρόεδρο. Πολλά μπορούμε να συζητήσουμε εδώ μεταξύ μα. Και εγώ να το συζητήσω μαζί σα ευχαρίστω. Αλλά α υπάρχει ο χρόνο για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, έχετε δίκιο, λέει ο πρόεδρο. Είμαστε δύο μήκο κύματο. Και τον κύριο Ζήμων. Το ΕΛΚΑ με τους κυρίους Φάρμπερ και Χοκμάρκ το, η, η πράσινη με τον κύριο Λάμπερτς η Γκουε με τον κύριο Ντεμάζη που δυστυχώς λείπει και οι σοσιαλιστές με τον υποφυνόμενο αναφέρονται στο πακέτο για τον περιορισμό του κινδύνου με στόχο πραγματικά σε όλους τους τομείς να περιοριστεί ο κίνδυνος, όχι να δημιουργηθεί περιττέρω κίνδυνος και αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Θέλω να υπενθυμίσω και να τονίσω ότι η αναλογικότητα για μένα είναι νοητή και προς τις δύο κατευθύνσεις και προς τα άνω, εκεί δηλαδή που είναι υψηλότερος ο κίνδυνος και άρα χρειάζεται περισσότερη επαγρύπνηση και εποπτεία και αναλογικότητα προς τα κάτω όπου μπορεί ένα κριτήριο ε, ελάφρυνσης της επαγρύπνησης να είναι μεγαλύτερη κρατική συμμετοχή στην διαμόρφωση του χρέους. Αλλά βεβαίως πολύ ευχαρίστω, όπως είπε και ο κύριος Φέρμπερ, να συζητήσουμε όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν ακουστεί από πολλές πλευρές και που έχουν όλες την αξία τους, γιατί ορίζουν ποιοτικά το πότε μία τράπεζα δεν πρέπει να υπάγεται σε αυτή την αυστηρή ε, νομοθεσία. Αυτά είναι τα θέματα που θα μας απασχολούν στις επόμενες εβδομάδες μέχρι την κατάρτιση της έκθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας προσφέρατε πολύ food for thought. Ευχαριστώ. Thank you very much. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε όσον αφορά τα θέματα πέραν του fast track, έχουμε το χρονοδιάγραμμα 11 Εβδόμου θα γίνει η συζήτηση. Σεπτέμβριο. 7 Σεπτεμβρίου οι τροπολογίε είναι η τελική ημερομηνία. 16 και 19 θα συζητήσουμε τι τροπολογίε. Ψήφιση τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Για το fast track όπως ήδη αποφασίσαμε ακόμη δεν έχουμε το χρονοδιάγραμμα αλλά για να υπάρξει περιθώριο για τους τριμερείς διαλόγους. Να αρχίσουμε τον Σεπτέμβριο. Άρα θα πρέπει να έχουμε το σχέδιο της έκθεσης το αργότερο τέλη Μαΐου. Αυτό το καταλάβουν όλοι. Πρέπει. Οπότε ο Γκουνάρ να έχει την δυνατότητα να προχωρήσουμε όχι στα τυφλά με το fast tracking Άρα θα πρέπει να δίνει και άλλη προσπάθεια. Δηλαδή θα πρέπει να, ληφθεί, να ληφθούν υπόψη όλες οι εξελίξεις. Οπότε να επανέλθουμε στο fast track όταν τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα και θα έχουμε τα βασικά στοιχεία που αναφέρατε. Όχι, αυτό δεν θα κρυθεί σήμερα. Οπότε κατάλαβα πού το πας. Ότι δηλαδή χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και άλλες μεταβλητές. Και έτσι να προχωρήσουμε κάποια συνέπεια και συγκρότηση για το fast tracking. Αλλά προς το παρόν έχουμε μόνο μία σχετική απόφαση που έχει συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας. Τώρα. Στον έλεγχο. Α, διακόπτει ο κύριο Χόκμαρ. Έχουμε την απόφαση των ε, συντονιστών δεδομένη. Ναι, ναι, λέει ο πρόεδρος. Αποφασίστηκε να μην προχωρήσουμε και να επανέλθουμε όμως στο θέμα του φαστάκινγκ πριν τις θερινές διακοπές. Ακριβώς για το λόγο που είπες κι εσύ. Κάτι λέει ο κύριος Μπάλτς εκτός μικροφώνου. Ναι, ναι, όποτε πρέπει ε, σε αυτά είμαστε IT. Α, περιβάλλον σου έχεις το λόγο. Τώρα παρεμπιπτόντως να πω τα εξή ότι εάν η Επιτροπή πρότεινε αυτή την τροπολογία των BRD σε χωριστό φάκελο, αυτό είναι θέμα της Επιτροπής μας σε πλήρη σύνθεση να αποφασιστεί η τύχη αυτή τη πρόταση. Οπότε, αν αποφασίσουμε να κάνουμε το fast track ή όχι για αυτή την πρόταση, από πλευρά νομοθετική, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το κρίνουν οι συντονιστέ. Και το στον μετά από συζήτηση, η διαπραγματευτική ομάδα και να μην ξανανοίξει το θέμα στην Επιτροπή σε πλήρη σύνθεση. Αλλά ας το δούμε προσεκτικά ακριβώς με το πνεύμα που μας εξήγησε ο εισηγητής. Και φυσικά να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι το θέμα θα πρέπει να ξανανοίξει. Ευχαριστώ. Επόμενο σημείο. Εδώ που κάνουμε τον έλεγχο, ο Μάρκους θα ασχοληθεί με το πρώτο μέρος. Μετά θα έχουμε έλλειψη αντιπροέδρου ε, εκτός αν έρθει κάποιος, γιατί έχουμε μια συνάντηση σημαντική τώρα. Ελπίζω σε κάνα μισά ώρα να επιστρέψω. good morning everybody. Καλημέρα σε όλους. We come to our scrutiny of uh, delegated... Λοιπόν, εξετάζουμε κατεξοδότηση πράξη εφαρμοστικά μέτρα. Έχουμε τρία μέτρα του επίπεδου 2 όσον αφορά τον κανονισμό για τους, για τους φορείς αξιολόγησης από την GD Φίσμα, η κυρία Σαλίφσκα. Ε, έσμα, ο κ. Βαλτζούγκ, Σωστά τα λέτε ονόματα. Ποιο θα ξεκινήσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Τσαλίφσκα, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. First of Καταρχάς, σας ευχαριστήσω πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσω με θυμόν το έργο μας όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού περί των διαφόρων φορέων αξιολόγησης, πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οπότε θα έρθω μέσω στην ουσία του θέματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την εντολή από τον κανονισμό να υιοθετήσει κάποιων μέτρων επίπεδου 2 όπως αποκαλούνται και να συντάξει εκθέσεις. Να σας πω με τα ότι όλες οι εντολές που μας δόθηκαν εκπληρώθηκαν. Κάναμε ό,τι ήταν αναγκαίο τον Οκτώβριο του 2016 μάλιστα. Υιοθετήσαμε τα εξής έγγραφα. Σεπτέμβριο του 2014. Τρεις ρυθμιστικές προδιαγραφές για την βάση, για την πλατφόρμα αξιολόγησης. Επίσης τα τέλη που επιβάλλουν στους πελάτες τους αυτοί οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης και μετά τα διάφορα, εξετάσαμε τα διάφορα θέματα διάθοσης. δομημένα εργαλεία για τις πιστώσεις. Τελειώσαμε λοιπόν τον Οκτώβριο του 2015 την έκθεση για το κατά πόσο χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση για την πιστοληπτική ε, ικανότητα και το 2016 τον Οκτώβριο υιοθετήσαμε έκθεση που αποτιμά την κατάσταση όσον αφορά την όλη αγορά ε, των οίκων αξιολόγηση και πόσο αποτελεσματικές είναι οι διάφορες διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό για αυτούς τους φορείς. Αυτή η έκθεση αναφέρεται ε, στις εντολές που προβλεπόταν για την υποβολή αναφορά στον κανονισμό. Όσον αφορά την έκθεση που θετήσαμε πέρσι. Να σας πω κάποια βασικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάναμε ανάλυση των στοιχείων, ήρθαμε σε επαφή με φορείς της αγοράς και πήραμε και απαντήσεις από την ΕΣΜΑ. Αναφερόμαστε στους βασικούς στόχους του κανονισμού στην έκθεσή μας. Πρώτο συμπέρασμα για την υπερβολική εξάρτηση από τους φορείς αξιολόγησης. Στην έκθεση διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το σύστημα αξιολόγησης. Μόνο συμπληρωματικά εργαλεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επενδυτέ να κάνουν την αξιολόγηση του κινδύνου και να αποφύγουν την εξάρτησή τους από αυτούς τους οίκους αξιολόγησης. Ενεθάρρυνε και ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του εποπτικούς φορεί να συνεχίσουν την προσπάθεια μείωσης μηχανιστικής εξάρτησης από τους οίκους αξιολόγησης, εξασφαλίζοντας ότι οι φορείς αγοράς χρησιμοποιούν συμπληρωματικά εργαλεία. Καθορίζει η έκθεση διάφορα εργαλεία προς χρήση. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε παρακολούθηση της κατάστασης που κρατεί στην αγορά και τις σχετικές, σχετικές μάλλον συγγνώμη, εξελίξεις όσον αφορά τον ανταγωνισμό που επικρατεί. Παρά τα αριθμιστικά μέτρα, η αγορά είναι πολύ συγκεντρωμένη. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη φύση της αγοράς, που είναι, προσφορά, ε, είναι αγορά προσφοράς και ζήτησης. Υπάρχει μεγάλη, μεγάλος σχετισμός ζήτησης και προσφοράς. Οι φορεί χρησιμοποιούν τους οίκου αξιολόγηση που αναγνωρίζονται από τους περισσότερου επενδυτέ. και οι επενδύτε προτιμούν να χρησιμοποιήσουν του οίκου αξιολόγηση εκείνους που τους προσφέρουν τη μεγαλύτερη κάλυψη για τα προϊόντα που ενδιαφέρονται. Παρακολουθούμε συνεχώς την αγορά. Αλλά Ίσως είναι δύσκολο να αλλάξει κάπως η κατάσταση. Όμως, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τυχόν φραγμούς για την είσοδο στην αγορά. Πρόσφατα τροποποίησαμε το σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών για τη χαρτογράφηση των οίκων αξιολόγησης που πρότειναν οι διάφοροι αρμόδιοι φορείς. Αυτή η τροποποίηση που επιφέραμε είχε σκοπό να εξασφαλίσει ισότιμη αντιμετώπιση της βαθμολόγησης των οίκων αξιολόγησης ανεξάρτητα από το μέγεθος. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε την ευρύτερη αποδοχή και των μικρότερων φορέων αξιολόγησης. Κάτι άλλο, πάρα πολύ σημαντικό, που είναι στόχος του κανονισμού, ε, δηλαδή σύγκρουση συμφερόντων και σωστή διακυβέρνηση του συστήματος, τα εθετηθέντα μέτρα πιστεύουμε ότι έχουν προληπτικό χαρακτήρα κυρίως και πρέπει να συμβάλλουν κανονικά στην αυξανόμενη ανεξαρτησία των διαφόρων φορέων. Και έτσι η ΕΣΜΑ μέσω των μέτρων αυτών μπορεί να εξασφαλίζει ότι οι οίκοι αξιολόγησης που κινούνται στην αγορά πληρούν τα κριτήρια, τα αναγκαία. Όμως, τι παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την αναλογικότητα κάποιων μέτρων. Κυρίως όσον αφορά τις κυρώσεις. Ε, συγκρίση με το τζίρο των οίκων αξιολόγησης. Βλέπουμε δυσαναλογία μεταξύ ε, φορέων αξιολόγηση που είναι μεγάλη και εκείνο που είναι μικρή. Άρα προβαίνουμε σε περαιτέρω ανάλυση της αγοράς. Επιτηρούμε την αγορά και να δούμε κατά πόσον έχουν σωστά αποτελέσματα αυτά τα μέτρα όσον αφορά τα διαθρωμένα μέσα χρηματοδότησης. Συμπεράναμε το 2016 ότι είναι πολύ πρόημο να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο του κανονισμού τώρα. Κάποιες διατάξεις βλέπετε δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη. Άρα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην αγορά. Τέλος, όσον αφορά το κατά πόσο να έχουμε ευρωπαϊκή αξιολόγηση για το κρατικό χρέος δεν χρειάζεται τώρα να έχουμε ευρωπαϊκό φορέα αξιολόγησης που ασχολείται κυρίως με το κρατικό χρέος κατά την άποψή μας κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει αύξηση του κόστους και δεν θα δώσει τόσο μεγάλη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην αγορά. Και τίθεται και το θέμα τη ανεξαρτησία ενό φορέα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Και πώ θα γίνει αντιληπτό αυτό ο φορέα από επενδυτέ εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ποιο είναι το γενικό συμπέρασμα. Αναφέρει λοιπόν η έκθεση στα πορίσματά τη ότι ο κανονισμό και τα νέα μέτρα θα έπρεπε να έχουν θετικό μακροπρόθεσμο ε, αντίκτυπο όσον αφορά την αγορά των οίκων αξιολόγηση. Χρειάζεται χρόνο όμω να δούμε ποιο θα είναι ο πλήρη ε, αντίκτυπο, τα πλήρη αποτελέσματα των μέτρων. Εν κατακλείδη, αυτά είναι τα βασικά απορίσματα της εκθέσεως. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με την ΕΣΜΑ θα συνεχίσει τις προσπάθειες θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και πριν υιοθετηθούν περαιτέρω μέτρα, αυτό θα κάνουμε. Για την ώρα λοιπόν συνεχίζουμε την σε εποπτεία της αγοράς και μάλιστα και σε στενή συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα και είμαι έτοιμη να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Η ΕΣΜΑ. Ο κ. Φανβάλζουμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ την Επιτροπή σας που οργάνωσε αυτού του είδους την ε, συνάντηση για τον ε, έλεγχο όσον αφορά ε, τον κανονισμό για τις εταιρείες αυτές αξιολόγησης και να σας πω ότι τι βρήκαμε, τι έχουμε διαπιστώσει μέσα από την ε, δουλειά μας όσον αφορά αυτά τα σημαντικά θέματα. Πρώτα πρώτα να σας πω ποιο είναι το πλαίσιο αυτού του κανονισμού CRA, αυτές τις εταιρείε δηλαδή, στο επίπεδο 2. Και κατόπιν να δούμε τι ισχύει όσον αφορά το CRA 3 και τέλος να συζητήσουμε στο τι θα ακολουθήσουμε σαν ρότα πολιτική στο μέλλον. Πρώτα-πρώτα να σας πω πώς έχει το ευρύτερο τοπίο όσον αφορά της εταιρείας επιστολικής αξιολόγησης και το νομικό σχετικό πλαίσιο για τη δουλειά μας. Ο κανονισμός ε, θεσπής του 2009 ήταν κάτι που το να γίνει γιατί για πρώτη φορά θα είχαμε αυτό το πλαίσιο εποπτείας για αυτού του είδους τόσο σημαντικούς παίκτες της ε, ε, χρηματαγορές και πρόκειτο επίσης για κάτι πάρα πολύ βασικό για να αντιμετωπίσουμε τα ίδια της κρίσης του 2008 και αυτό ε, έπαιξε σημαντικό ρόλο και συνεχίζει να παίξει σημαντικό ρόλο σε την προστασία του, ε, του επενδυτή, τη σταθερότητα της αγοράς και την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η ΕΣΜΑ μπήκε λοιπόν στη σκηνή με αυτόν τον κανονισμό υπαριθμών 2 και ήταν η μόνη υποπτική αρχή για αυτές τις εταιρείες το 2011. Σε αυτή την πρώτη φάση η να έχουμε να είμαστε μάλλον αξιόπιστος και αποτελεσματικός επόπτης όσον αφορά αυτές τις εταιρείε όσες λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτά τα μέτρα είπαμε ότι θα προσέξουμε τι γίνεται όσον αφορά ε, την δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων τους όσο αφορά τα πρότυπα υποπτίας που ήταν σημαντικά και τώρα με τον κανονισμό με το CRA 3 το, του 13 ε, ε, εξελίσσουμε τη δουλειά μας και επίσης ε, μας ζήτησαν να έχουμε κάποιους τεχνικά πρότυπα ούτω ώστε να υπάρχουν κάποιες ε, πλατφόρμες ε, πληροφορική που να είναι πιο φιλόδοξες, πιο καινοτόμε, και έτσι να έχουν περισσότερη διαφάνεια αλλά και προστασία του καναλωτή και τώρα μπορώ να πω κάνοντας αναδρομή στα τελευταία τέσσερα χρόνια ότι ό,τι μας ζητήσανε το πετύχαμε. Τώρα, όσον αφορά όλα αυτά τα τεχνικά πρότυπα, αυτό ίσως που είναι πιο αισθητό στον εξωτερικό παρατηρητή είναι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αξιολόγησης που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2016 και έχουμε ένα website και τώρα εκεί πέρα έχουμε ολόκληρο πόρτα, ολόκληρη ε, τέτοια θύρα, πύλη τέλος πάντων ε, και κάποιος μπορεί εκεί να δουλέψει δωρεάν και χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει αλλού και είπαμε ότι έτσι υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα των εταιριών αυτών και έτσι κάτι γίνεται πιο απλό ενώ πριν ήταν κάτι δαπανηρό και μπλεγμένο για τους ε, επενδυτές Επίσης κάτι άλλο είναι το τι χρεώνουν για τις υπηρεσίες τους στους πελάτες αυτές οι εταιρείε. Τώρα συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια υποπτία για αυτά που χρεώνουν για τη δουλειά τους αυτές οι εταιρείε, να μην έχουμε πρακτικές δυσμενούς διάκρισης και να ισχύει θεμητός συνταγωνισμό και να μην έχουμε και συγκρούσεις συμφερόντων. Ε, πέραν τώρα των τεχνικών προτύπων για το CRE3 ε, έχουμε αυτή την πλατφόρμα για διάφορα δύσκολα πράγματα όπως αυτή η αγορά και για το κατά πόσον είναι βιώσιμες αυτές οι αξιολογήσεις. Να μην επιστρέψουμε τώρα ε, στις λεπτομέρειες, αλλά να, δούμε ποια είναι τα σημαντικά σημεία. Όσον αφορά την υπερβολική στήριξη σε αυτού του είδους αξιολογήσεις, όπως είπαμε, θα είναι δύσκολο να καλύψουμε όλο αυτό το θέμα γιατί έχουμε πολλά σημαντικά νομοθετήματα στο κοινωτικό δίκαιο που παραπέμπουν στην ε, πιστοληπτική αξιολόγηση. Επίση, είναι σημαντικό να δούμε το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ αυτέ οι εταιρείε για αυτού που δεν έχουν ε, για να επενδύσουν ε, εναλλακτικέ. Και για αυτό το λόγο είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει λιγότερη εξάρτηση από αυτές τις εταιρείες και όχι να, τις, να καταργήσουμε τελείως την χρήση τους και γι' αυτό και ε, στην έμπα και στην ΑΙΟΠΑ συνεργαστήκαμε πάρα πολύ, ώστε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες άρτιες τεχνικές εποπτικές ε, και όλα αυτά δημοσιοποιήθηκαν το 2016. Επίσης όσον αφορά τις τεχνικές συμβουλές για ανταγωνισμό κλπ. Ε, είδαμε ότι παρά κάποιες πρωτοβουλίες του CRA3 η αγορά των εταιριών αυτών γνωρίζει συγκέντρωση. δηλαδή έχουμε τρεις-τέσσερις εταιρείε που κυριαρχούν. Εμεί θα συνεχίσουμε να πασχίζουμε το ώστε να ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμό και όλα να λειτουργούν ε, ε, εύρυθμα. Πρόσφατα είχαμε κάποιο είδου ε, ενημέρωση και προσπαθήσαμε να πάμε προς μια αναρμοσμένη προσέγγιση και να δούμε πώς μπορεί να μπουν στο παιχνίδι και μικρότερες τέτοιες εταιρείες. Επίσης, επισύρω την προσοχή σας στο ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα στις αρμοδιότητες για κυρώσεις που έχουμε. Και αυτό θα πρέπει όμως να το εξελίξουμε και να υπάρχει περισσότερη αναλογικότητα και να υπάρχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Αλλά αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με αυτά τα οποία επιτάσσει ο κανονισμός CRA και τα πρόστιμα να έχουν σχέση και να εξαρτώνται από το τζίρο της κάθε εταιρεία. Άρα είναι σημαντικό να αυξηθεί η αξιοπιστία ε, του εποπτικού μας πλαισίου. Τέλος, θα ήθελα να σας θίξω θέμα ε, που αφορά το θέμα του, του, του, του μέλλοντος, γιατί όπως θα είδατε τον περασμένο μήνα είχαμε αυτό το έγγραφο διαβούλευση όσον αφορά τις κατευθυντήριες για ε, ε, αυτό το καθεστώς των εταιριών, δηλαδή το πώς θα επιτρέπονται ε, αξιολογήσεις πιστοληπτικές που θα προέρχονται από εταιρεία τρίτης χώρας και είπαμε ότι έχουμε πολλές τέτοιες οπότε χρειάζεται μέχρι τον Ιούνιο του 2018 να έχουμε αναθεωρήσει το τι ισχύει για να συνεχίσουν να ισχύουν τα υψηλά πρότυπα των αξιολογήσεων όπως επιτάσσονται από τον κανονισμό και όπως προσδοκά η, η ΕΣΜΑ. Εγκατακλείδη σα ευχαριστώ για την διαφορετική στη δουλειά μα και για τον κονισμό μα και θα συνεχίσουμε το, το, το καθήκον μα το εποπτικό να εξασφαλίσουμε προστασία υψηλού επίπεδου για του ε, ε επενδυτέ, για του χρήστε των αξιολογήσεων, σταθερότητα στην αγορά και εύρυθμη λειτουργία τη αγορά και για το έργο μα. Θα χρησιμοποιήσουμε την ε, εμπειρία μας, όλα τα εργαλεία πολιτικής που υπάρχουν και επίσης θα προτείνουμε την αναθεώρηση των ε, ισχυών των ε, Ό,τι ερωτήσει έχετε θα απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ και σας ακούσουμε τώρα τον Πολ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και την Επιτροπή και την ΕΣΜΑ που είναι εδώ. Ευχαριστώ για όλη την καλή δουλειά. Είναι βέβαια φύση αυτής της δουλειάς που γίνεται ή που δεν έχει γίνει. Και του τουλεχθέντος πρέπει να κοιτάξουμε και τη δουλειά που δεν έχει γίνει. Διότι εγώ αισθάνομαι μεγάλη δυσφορία εδώ, καθώς μάλιστα λέει η Επιτροπή ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Γιατί βλέπουμε προβλήματα, μεγάλη συγκέντρωση, τρεις επιχειρήσεις με το 90 και μάλιστα αμερικανικές επιχειρήσεις. Αλλαγή δεν υπάρχει, ούτε και αναμένεται. Και αν αυτό το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι μικρές CRAs έρχονται και μας λένε ότι η ECB παρεμποδίζει την είσοδό τους, ε, τι να πούμε τότε, δεν μπορούμε να περιμένουμε ε, αδρανείς τις εξελίξεις. Να σας πω εγώ ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Θα επικρατήσουν οι τρεις αυτές επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια. Και περιμένω επίσης ανταγωνισμό, διαφοροποίηση, περισσότερες εισόδους, μεγαλύτερη ποικιλία και διαφοροποίηση και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η Επιτροπή ούτως επίν άνευ εταίρου απορρίπτει την ιδέα μιας ε, υπηρεσίας που θα έλεγχε την κατάσταση που δεν θα είχε δηλαδή στόχο το κέρδος και έτσι θα επέτρεπε μια ρύθμιση. Γιατί λοιπόν όχι. Και γιατί η ΣΥΒΗ ε, παρεμποδίζει την είσοδο μικρών επιχειρήσεων χρηματοπιστωτικής αξιολόγησης. Επίσης, κάτι άλλο που με προβληματίζει ιδιαίτερος είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπει εναλλακτικές να υπάρχουν, αλλά δεν τις έχει υιοθετήσει η Επιτροπή. Όπως έχουμε στο STS, στο CR, την ε, μεγάλη εξάρτηση που διαπιστώνουμε και το κοινοβούλιο σας λέει ας αλλάξουμε την ιεράρχηση των μεθόδων. Μια τυποποιημένη προσέγγιση ας είναι ιεραρχικά προτιμότερη από την εξωτερική αξιολόγηση. Δεύτερον, δεν υπάρχει αξιολόγηση, λέτε, για τα ε, δομημένα. Ε, το Κοινοβούλιο τώρα με τον ε, φάκελο SDS σας λέει ότι μπορεί να υπάρχει μια εποπτεία και κρίσιμο είναι να έχουμε στη θέση μας τα στοιχεία που χρειάζονται για τα πολύ περίπλοκα δομημένα προϊόντα. Και ναι, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά εναλλακτικέ επίσης υπάρχουν. Και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο υποστηρίζει αυτές τις προσεγγίσεις. Επτά από τις 41 CRA επίσης έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η εικόνα στο προσεχές διάστημα, διάστημα και εν ώψη της συγκέντρωσης αλλά και όταν έρθει η ώρα να υπάρχουν ακόμα CRA στο Λονδίνο αλλά να μην υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ο μιλητής εκ μέρους των ομάδων, η κυρία Κάινεν πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Αντίθετα από τις επικρίσεις που ακούστηκαν μόλις τώρα, θέλω να πω ότι αισθάνομαι αρκετά ικανοποιημένη από τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα η Επιτροπή στον τομέα αυτών. Σημερίζομαι αρκετά από τα προβλήματα που διαπιστώνουμε σε σχέση με τη CRA και την νομοθεσία. Πρώτον, ε, πολύ έντονη συγκέντρωση της αγορά, στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα δεν βλέπω τι θα εξυπηρετούσε μια δημόσια υπηρεσία αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας εκτός από το να εξαρτάται πάρα πολύ από τη λεγόμενη κοινή γνώμη πέραν των κακών προθέσεων, γιατί φαντάζομαι ότι και οι πολύ καλές προθέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ κακά αποτελέσματα ή να μας παραπλανήσουν. Μία δημόσια αρχή πιστοποιητικής ε, αξιολόγησης είναι λίγο σαν την ε, πρόβλεψη της μετεωρολογικής, γιατί μπορεί καλής να έχει καλή μεθοδολογία και καλές προθέσεις, αλλά πάλι δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί. Άρα το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλή εποπτεία. Διαφάνεια και ποιότητα στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Και μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα όταν χρησιμοποιηθεί και αναπτυχθεί, όταν αναπτυχθεί, μπορεί να αξιοποιηθεί πιστεύω και για να εξασφαλιστεί η συγκριτικότητα, η συγκρισιμότητα και μια διαφορετική ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας και βεβαίως εγώ θα ήθελα να έχω μια μεγαλύτερη ποικιλία ως προς την ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας γιατί είναι τεράστιος ο κίνδυνος αν δούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε αντικειμενική αξιολόγηση. Η συγκέντρωση λοιπόν στην αγορά είναι τεράστιο πρόβλημα. Θα ήταν καλύτερο να έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στην ευρωπαϊκών αλλά από την άλλη είναι και μια δουλειά πολύ απαιτητική με πολύ μεγάλη επιβάρυνση κόστους και άρα δεν είναι πιθανό εύκολα να αναδυθούν τέτοιες επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη όπως άλλωστε συνέβη και με το τραπεζικό τομέα. Έτσι λοιπόν θέλω να ακούσω πώς λειτουργεί η εποπτεία μας, φαίνεται να λειτουργεί ικανοποιητικά, αλλά στην διαχείριση και βέβαια τα, ε, τις κρυφές συγκρούσεις συμφερόντων, πώς λειτουργεί. Και εγώ αναφέρομαι εδώ και στις αθέλητες ακόμη μεροληπτικές επιλογές, αθέλητα μεροληπτικές επιλογές, όχι τις εσκεμμένες. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό να εστιαστεί στο μέλλον η ΕΣΜΑ. Και μια και υπάρχει συγκέντρωση στην αγορά, κατά πάσα πιθανότητα στο μέλλον θα εξαρτηθούμε ακόμα περισσότερο από τις εξωτερικές αξιολογήσεις. Για να υπάρχει ένα, μια, μια υψηλού επίπεδου εποπτεία. Έτσι λοιπόν θέλουμε να δούμε κάποια πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για το μέλλον, ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι στο επίπεδο, δεν είναι στο επίκεντρο της ε, μελέτης τώρα. Είναι αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων, ε, ε, αλλά και η συμπερίληψη φερρυπίν περιβαλλοντικών κινδύνων στην αξιολόγηση στο μέλλον, που δεν ρυθμίζει αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια νομοθεσία. και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει αυτά τα θέματα να τα συμπεριλάβει στο έργο της, στο μέλλον για την αξιολόγηση ποιότητα, ζητήματα διακυβέρνησης ή και δευτεροβάθμια αρτίες στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. ECR, Ashley Fox. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ξεκίνησα τη δουλειά μου για τα CRS, ήμουν τον κύριο Γκοζές και τον κύριο Ντομίνιτσι. Ήταν από τα πρώτα χαρτοφυλάκια που ανέλαβα όταν εξελέγει το 2009 για τους οίκους αξιολόγησης. Και οι στόχοι έκτοτε του Κοινοβουλίου δεν άλλαξαν. Θέλαμε να αυξήσουμε τη διαφάνεια και να μειώσουμε τις πιθανότητε συγκρούσεων συμφερόντων. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΣΜΑ για τι παρουσιάσει τους. Οι κανονισμοί που μέχρι τώρα εγκρίναμε βοήθησαν την επίτευξη αυτών. Θέλαμε επίσης να μειώσουμε την εξάρτηση από τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ε, δυνατότητας ε, και τα πετύχαμε όλα. Δεν πρέπει να είμαστε έκπληκτοι. Δεν είναι δυνατόν να θεσπίζουμε κανονισμούς και οδηγίες από εδώ και να περιμένουμε ξαφνικά ε, να έχουμε πολλές ε, νέες εταιρείες να μπαίνουν και η αγορά να εξαρτάται λιγότερα, λιγότερο από τις αξιολογήσεις. Κυρίως όταν το κάνουμε εμείς εδώ, στο Κοινοβούλιο. Διότι τότε που ήμουν ασκιώδης για το CRA 3, που θεσπίζαμε νομοθεσία για τη μείωση τη εξάρτηση, τότε ήμουν και σκιώδη για το Solvency 2. Και τι θεσπίζαμε σε νομοθεσία. Ότι διάφορα ιδρύματα θα μπορούσαν να θεσπίζουν σε διάφορα μέσα με συγκεκριμένη αξιολόγηση, συγκεκριμένη βαθμολογία. Άρα, άμα θεσπίζουμε αντικρουόμενα πράγματα, έχουμε και αντικρουόμενα αποτελέσματα. Το είχα πει, αλλά επιματέω. Τόσον αφορά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ζητώ το εξής να μου πει η ΕΣΜΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι αξιολόγηση κάνατε όσον αφορά την αύξηση του διοικητικού άχθους που συνεπάγεται η εφαρμογή του κανονισμού όσον αφορά τις εταιρείε αξιολόγησης διότι οι μεγάλες τρεις αμερικανικές εταιρείε που ανέφερε ο κύριος Τάγκ και οι οποίες δεν του αρέσουν είναι σε πολύ καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν το διοικητικό άχθος από ότι είναι ερχόμενες εταιρείε. Και τα μετά ευρωβουλευτές όταν έχουν επιβάλει αυτό το συμπληρωματικό διοικητικό άχθος στις νεοσερχόμενες, έχοντας κάνει αυτό, γιατί εξακολουθούν να ευημερούν οι τρεις μεγάλες εταιρείε. Εάν έγινε αξιολόγηση θα με ενδιαφέραν τη δω. Το διοικητικό άχθος που επέβαλαν συνάδελφοι στις εταιρείε αξιολόγησης ε, δυσχεραίνει την είσοδο νέων εταιρείων στην αγορά. Δεν εκπλήσωμε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκός φορέας αξιολόγησης. Το είχαμε πει από την αρχή, ο μόνος σκοπός τέτοιες υπηρεσίες θα ήταν να λέει στους επενδυτές πόσο καλό θα ήταν να επενδύσουν στο ελληνικό χρέος. Θα ήταν άσκηση πολιτικής και κανένας δεν θα έδινε την παραμικρή προσοχή σε αυτό. Αν ο κύριος Τάγκ, οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι φίλοι του θεωρούν ότι αυτό έχει αξία, τότε χρησιμοποιήστε τα δικά σας χρήματα αν δημιουργήσετε έναν φορέα αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα και να πείτε εσεί στου επενδυτέ πόσο καλό θα ήταν να επενδύσουν στο ελληνικό χρέο και να δείτε πόσο επιτυχεί θα είσαστε στην αγορά κάνοντά το αυτό. Θα είναι πλήρε χάσιμο χρόνου και ε, διασπάθηση δημοσίου χρήματο. Στο τελευταίο, το τελευταίο RTS εφαρμόστηκε 1η Πρώτου 2017. Άρα είναι πολύ πρόημο να κάνουμε μια αξιολόγηση. Να δούμε κατά πόσο ήταν επιτυχές ή όχι. Ανησυχώ λιγουλάκι, διότι τι διαβάζω. Ότι συζητείται θέσπιση σε περισσότερες νομοθεσίες όσον αφορά την έγκριση και υποστήριξη έχουμε πρόβλημα εδώ με τι υπερβολικές ρυθμίσει. Ποτέ δεν επιτρέπουμε στα χρηματοστατικά ιδρύματα μια περίοδο ηρεμία. Πάντα προσπαθούμε να αλλάζουμε κάτι για να μας βλέπουν ότι κάνουμε κάτι. Το είχαμε αυτό και στο προηγούμενο σημείο που συζητήσαμε, το CRR. Συνηθίζει κανείς με μια ομάδα κανονισμών, μιλώντα για τι τράπεζε τώρα, και μεταλλάζουμε πάλι του κανονισμού. Αφήστε ε, τι εταιρείε αξιολόγηση κάνα δύο χρόνια στην ησυχία του. Μην μπλεκόσαστε, μην μπερδεύεστε. Αφήστε του δύο-τρία χρόνια. Κάντε μια ήρεμη αξιολόγηση στο τέλο τη περίοδου αυτή και μετά. Κάντε μια αποτίμηση και να δείτε κατά πόσο χρειάζονται αλλαγέ. Η ΕΣΜΑ πάντα λέει πόσο σας λείπει το προσωπικό, λέτε χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους και άλλα χρήματα. Ε, ότι έχετε τους ευθύνε. Λοιπόν, μην κάνετε αυτό. Ηρεμήστε για κάνα δύο χρόνια. Ευχαριστώ. Αυτή η υπερβολική ρύθμιση δεν εμποδίζει τη δημιουργία νέων υπηρεσιών που πλασιάζονται. Άλτε. Ο συνάδελφος έχει το λόγο. Η συνάδελφος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΣΜΑ για την ανταλλαγή των απόψεων και αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΣΜΑ και ότι τα μέτρα επίπεδου 2 είναι όλα εφαρμοστέα. Να δούμε και κατά πόσο έχουμε πετύχει στη μεταρρύθμιση της αγοράς των οίκων αξιολόγησης. Όπως αναφέρθηκε θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για ανταγωνισμό στην αγορά αυτή. Ήταν βασικός μας στόχος και έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Βλέποντας το όλο σκηνικό μοιάζει με το πρωτάθλημα το Ολλανδικό. Πάντα μια από τι μεγάλες Φάιενορντ με Άγιαξ και λοιπά, η Φάιενορντ ή ο Άγιαξ νικούν. Πάντα μια από τις μεγάλες ομάδες. Εδώ φέτος ευτυχώς αγιαξ νικουν είναι πρωταθλήτρια. Σταματά φετος είναι προταλήτρια. Σταματάει η συζήτηση, διότι στο Ολλανδικό πρωτάθλημα είναι ακόμα δυνατόν και άλλη ομάδα να πάρει το κύπελο. Όπως η Βιτέσε το κυπελο οπως η πρόσφατα στη χώρα μας. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει στην αγορά των CRAs. Διότι έχουμε ένα λιγοπόλιο εκεί. 93% είναι στα χέρια των τριών μεγάλων εταιριών και υπάρχουν πολλοί νέοι ερχόμενοι, αλλά οι εταιρείε αυτές παραμένουν πάρα πολύ μικρές. Ένας φραγμός για μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των καταχωρημένων CRAs δεν αναγνωρίζονται σαν εξωτερικές υπηρεσίες αξιολογήσεως. Στην περίπτωση του DBRS, του Καναδικού Φορέα, ε, εκεί ε, τα μέτρα επέτρεψαν μεγαλύτερη προς την αγορά. Ήθελα να το παρακολουθήσει το θέμα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ερώτησή μας είναι, η ΕΣΜΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συζητήσατε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το θέμα αυτό. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των συζητήσεων, υπάρχουν συμπεράσματα. Δεύτερη ερώτηση οι τροπολογίες του κανονισμού που έγινε το 2013. Στο άρθρο 8 Δέλτα προβλέπεται η απέτηση να πρέπει να διορίζεται και δεύτερος φορέας για κάποια έκδοση. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τι εταιρείε που έχουν λιγότερο 10% τη αγορά. Στην έκθεση του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι είναι πάρα πολύ προήμο να προβούν σε μια αξιολόγηση τη διάταξη. Επίση, συνεπέρανε ότι δεν έχει εφαρμοστεί το μέτρο πλήρω σε εθνικό επίπεδο. Τώρα πέρασε άλλο ένα εξάμεινο. Ποια είναι η εξολόγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει εφαρμοστεί πλήρω η διάταξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εθελοντική μορφή τη διάταξης δεν καλύπτει επαρκώς τις μικρές εταιρείες. Μήπως γίνεται υποκειμενική αξιολόγηση των κριτηρίων. Και τι θεωρείται αποδοχή από πλευρά πιστωτών αντικειμενικά. Η έκθεση του Οκτωβρίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι έλεγε ότι οι κυρώσει σε περίπτωση συγκρούσεων συμφερόντων δεν έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα οι ε, Το έχετε εξετάσει εν τω μεταξύ περαιτέρω το θέμα, είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε η ΕΣΜΑ. Για τους πρασίνους τώρα λέει ο Πρόεδρος. κυρία Μαρίζα Ματίας, αλλά δεν παρίσταται. Υπάρχει άλλος για την αριστερά, όχι. Άρα πάμε στους πρασίνους. Σβέν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριο Γκίκολτ. Και εγώ θυμάμαι πολύ καλά τις συζητήσεις τότε που είπε ο συνάδελφος που ξεκίνησε το 2009 και θέλω να σας πω ότι είναι ξεκάθαρη η στόχη μας. Άρα τώρα είναι θεμητό κάποιος να ζυγίσει το τι πέτυχε και τι όχι. Δεν είναι σαφές. Θέλει περισσότερο ανταγωνισμό, περισσότερους παίκτες στην αγορά. Άρα θεμητά κανείς προβληματίζεται. Ακριβώς όπως έχει ρυθμιστεί και στο νόμο. Αγαπητέ συνάδελφε Fox, εμείς ποτέ δεν θέλαμε να υπάρχουν δημόσιε εταιρείε αξιολόγηση. Σας παραπέμπω στη ζήτησή μας. Γι' αυτό λέμε για ίδρυμα το οποίο πολιτικά να είναι ουδέτερο. Φοβόμαστε όπως και εσύ ότι εάν υπάρχει τέτοιο ίδρυμα θα υφίσταται πίεση και άρα δεν θα είναι αξιολογήσεις αυθεντικές έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το τι εναλλακτικές θα μπορούσαν να υπάρξουν. Και υπάρχει ενδιάμεση λύση μεταξύ δημόσιας εταιρεία και από την άλλη μεριά του ολιγοπολίου που τώρα ισχύει. Έχουμε νέους ε, παίκτες, ιδιώτες. που μπορούν να σταθούν. Και γίνεται να υπάρχει ένα διαφορετικό σύστημα, ούτω ώστε να υπάρχουν θεσμικές, κανονιστικές τέλο πάντων αξιολογήσεις. Και αυτό μπορεί να γίνει από έναν φορέα αξιολόγησης και έτσι οι μικρότεροι παίκτες να μπορούν να συμμετάσχουν. Αλλά και, και τα εκδούντα, οι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ξεφύγουν από το, από το λιγοπόλιο. Υπάρχουν σημαντικέ ενδιαφέρουσες έρευνες και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετήσατε εκείνες τι προτάσει. Τα λάβατε υπόψη. Άλλη ερώτηση. Με τον Άσπλη Φόξ συμφωνώ σε ένα σημείο ότι θα πρέπει τη σήμερα ημέρα να ρίξουμε περισσότερους πόρους, περισσότερες ε, προσπάθειες όσον αφορά την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων. Και τότε είχαμε πει ότι υπήρχε το 8β το και όσον αφορά την ενημέρωση για κάποιο είδους ε, δομημένα χρηματοπιστωτικά εργαλεία για διάφορα τέτοια περίπλοκα εργαλεία να υπήρχε αυτό το σύστημα τόσο ώστε να είναι ευκολότερο οι νέοι παίκτες στην αγορά να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Υπάρχει βάση δεδομένων. Τι κάνατε γι' αυτό για να εξασφαλίσετε την εφαρμογή του 8B. Μπορείτε να μας πείτε τι ισχύει. Τι κάνατε να εξασφαλίσετε ότι αυτά τα οποία θεσπίσαμε εφαρμόζονται. Εάν δεν εφαρμόζονται, πέστε μας πότε θα εξασφαλίσετε την εφαρμογή του δικαίου. Και Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Έχω και εγώ βάλει το όνομά μου στον κατάλογο για το Catch Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο συνάδελφο θέλει να μιλήσει. Ε, λοιπόν, εντάξει, Ας κουράσω λίγο ακόμα τους προσκεκλημένους μας με την ερώτηση αυτή. Θα έχετε αρκετό χρόνο για να απαντήσετε. Και πιάνομαι από τις ερωτήσεις ε, που είχε διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και ο κύριος Στάνκ. Αφήνω κατά μέρο το θέμα του ανταγωνισμού, που προφανώς ο στόχος δεν επιτυγχάνεται και δεν μπορούμε να είμαστε και ικανοποιημένοι από αυτήν την κατάσταση, το είπατε κι εσείς, αλλά πέραν αυτού για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία το Κοινοβούλιο είχε επιμείνει να συμπεριληφθούν ε, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στην αξιολόγηση, ε, στη μεθοδολογία αξιολόγησης. Τι έχει γίνει αυτό? Ε, το θέμα, δεδομένου ότι έχει όλο και πιο καυτή επικαιρότητα. Και επίσης θα προσθέσω ότι εάν τώρα γράφαμε την νομοθεσία θα προσθέταμε και την υποχρέωση παρακολούθησης της ποιότητας των φορολογικών δηλώσεων των ε, επιχειρήσεων και μάλιστα δεν νομίζω ότι μας εμποδίζει τίποτα μέσα στις κατευθυντήριες γραμμές και την αναθεώρησή τους να επισημάνουμε ιδιαίτερως την ε, ε, φορολογική αξιοπιστία και πρακτικές. Επίσης, ε, στις ε, διάφορες ανισχύσεις που εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιλαμβανόταν και το πώς οι αρχές αξιολόγησης παρενέβαιναν σε σχέση με πολιτικές διαδικασίες ή διαβουλεύσεις με την δράση τους και μάλιστα με κατάπληξη διαπίστωσα ότι η Standard Poor είχε κάνει παρέμβαση σε σχέση με την αξιοπιστία υποψηφίων στην εκλογική διαδικασία της Γαλλίας για τις προεδρικές εκλογές προβλέποντας νίκη του κυρίου Φιγιόν ή, ή του κυρίου Μακρόν. Επίσης. Το μοντέλο που εκφράζει η διαδικασία endorsement για τις αρχές αξιολόγησης πιστοληπτικής ε, ικανότητας. Είναι ένα μέσον για το μέλλον πιστεύω απαραίτητο και χρήσιμο να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του Brexit. Αυτό πιο πολύ προς την Επιτροπή. Έχετε αναλογιστεί τι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την καταχώρηση ως μέσο και όχι μόνο αρχές αξιολόγησης. Και τώρα που σας έχουμε γεμίσει το πιάτο και το μενού, ο καθένας από 7 λεπτά και ρωτώ ποιος θα λάβει πρώτος τον λόγο να ακολουθήσουμε την ίδια σειρά με την Επιτροπή πρώτη λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και πρέπει να πω ότι είναι πολλά τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Ε, εάν τυχόν και δεν μπορέσω να απαντήσω σε όλες σας ερωτήσεις, ε, παρακαλώ συγχωρήστε με. Θα δώσω απαντήσεις γραπτό στη συνέχεια. Ανταγωνισμός. Πολλές θέσεις εκφράστηκαν εδώ και νομίζω ότι αυτή είναι και η θέση της Επιτροπής λίγο πολύ. Δηλαδή ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι και προσπαθούμε να βρούμε λύση για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σε μεγάλο βαθμό βέβαια η αγορά υπαγορεύει τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, μπαίνουν σε αυτές τις ε, υπηρεσίες, στις αρχές αξιολόγησης και πιστοληπτικής ικανότητας διάφοροι παραγόντες, αλλά και πέραν του ότι πρέπει να αξιολογήσουμε στην κατάσταση, σημασία έχει η διαφάνεια, η ποιότητα, η διακυβέρνηση, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Και αυτό άλλωστε εξασφαλίζει και την ποιότητα της αξιολόγησης για τον επενδυτή και τον εκδότη. Η ένταξη λοιπόν στη είσοδο στην αγορά νέων υπηρεσιών, λέω, επιχειρήσεων αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα. Ε, θα μπορούσε να λάβει χώρα. Υπάρχουν πολλές μικρές όμως τέτοιες ε, αρχές αξιολόγησης, τις υποπτεύει ΕΣΜΑ. Βέβαια θα πρέπει καθεμιά να βρει την, ε, το δικό της μερίδιο αγοράς στη συνέχεια. Όπως και να έχει πρέπει να μελετήσουμε την αναλογικότητα ορισμένων μέτρων όπως κυρώσεις πολύ αυστηρές και βαριές σε σχέση με τον κύκλο οργανισμό των μικρών ε, αρχών αξιολόγησης και αμελητές σε σχέση με τον κύκλο εργασιών των μεγάλων. Άρα πρέπει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται κιόλα και σε αυτό προσπαθούμε στην Επιτροπή να βρούμε λύσεις βελτίωσης που δεν θα θέτουν αμφιβόλο και την ποιότητα της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, πράγμα πολύ σημαντικό βεβαίω που ήταν επίσης και στόχος ε, των κανονισμών. Στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά κριτήρια, δημοσιονομικές δηλώσεις, φορολογικές δηλώσεις, ε, μπορεί να απαντήσει ΕΣΜΑ πιστεύω, γιατί αυτά είναι και τα κριτήρια καταχώρησης ε, στην ε, υπηρεσία. Στην υπερβολική εξάρτηση από εξωτερικές αξιολογήσεις προτείνουμε στη, στις προτάσεις μας διαφορετικά εργαλεία τα οποία όμως σε ένα βαθμό μπορεί να είναι δαπανηρά για τον μεμονωμένο επενδυτή κύριος. Ακριβά πολύ που πάλι όμως προσφέρουν πρόσβαση σε πληροφορίες, την οποία προβλέπει και η πλατφόρμα. Άρα αυτή η διαφανής πρόσβαση σε πληροφορία προσφέρει περισσότερη πληροφόρηση για τον μεμονωμένο επενδυτή, αλλά ίσως να είναι όντως ακριβή αυτή η πληροφορία. Κεντρική τράπεζα. Ναι, γνωρίζουμε ότι κάποιοι μικροί φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θεωρούνται ε, σημαντικοί, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ξέρω ότι έχω γίνει συζητήσει των παρελθόν. Τώρα πια είναι η κατάσταση ακριβώς δεν το γνωρίζω, αλλά θα το σημειώσω για να ενημερωθώ λεπτομερέστερα. και θα μεταφερώ το θέμα αυτό βέβαια στην ιεραρχία μου ως ζήτημα που ενδιέφερε και πρέπει να παρακολουθήσουμε. Ε, πάντως ε, πάντα προσπαθούμε να ε, ευαισθητοποιούμε σε σχέση με το θέμα αυτό και να προάγουμε για όλα αυτά τα διαθέσιμα στην αγορά εργαλεία. Θα χρειαστεί να περάσει βέβαια κάποιος χρόνος καθώς είναι σχετικά νέα όλη αυτή η νομοθεσία, καινούρια. Κάποια μέτρα εφαρμόστηκαν μόλις από την αρχή του χρόνου, άρα είναι μέτρα καινούρια στην αγορά. Θα χρειαστούμε και εμείς κάποιο χρόνο λοιπόν για να διαπιστώσουμε την, τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών. Αλλά υπάρχουν ζητήματα όπως η αναλογικότητα των κυρώσεων που ήδη επεξεργαζόμαστε. Δεν ξέρω αν κάλυψα όλες τις ε, ερωτήσεις, ε, μάλλον όχι, αλλά πάντως ε, πολύ ευχαριστώ να τις καταγράψουμε και να απαντήσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Thank you, um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. questions. Let me first say... Λοιπόν, ποια είναι η πολιτική μας ε, δεν ασχολούμαστε τόσο με τον ανταγωνισμό. Εποπτεύουμε την αγορά λίγο πολύ. Τι πρέπει να απαντηθεί. Αν υπάρχει συγκέντρωση, υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση προφανώς. Γι' αυτό η ΕΣΜΑ εξετάζει κατά πολύ τις διαδικασίες βαθμολόγησης, την ποιότητα βαθμολογήσεως. και επί του προβλήματος της συγκέντρωσης. Γι' αυτό καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες και χρόνο εξετάζοντας τη κυβέρνηση των εταιριών αξιολόγησης και τους τρόπους ε, αξιολόγησης με ανεξάρτητο τρόπο. Θέλουμε να έχουμε μία βάση ποιοτική ανάλυση. Λαμβάνοντα υπόψη τη μεγάλη συγκέντρωση πάντα. Σε μια τέτοια αγορά με μεγάλη συγκέντρωση πρέπει να δούμε αν υπάρχουν νέε ερχόμενε εταιρείε. Είναι τέτοιο το βάρο για την είσοδο που είναι αδύνατο να μπουν στην αγορά. Βάσει στατιστικών στοιχείων δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν σε αυτή τη φάση 39 καταχωρημένες εταιρείες αξιολόγησης. Δύο-τρει νέε εταιρείε έρχονται στην αγορά το χρόνο κατά μέσο όρο. Όλε μικρομεσαίε εταιρείε αξιολόγηση. Άρα δεν είναι αδύνατον να εισέλθει στην αγορά μια καινούργια εταιρεία. το θέμα του endorsement, της έγκρισης και αναγνώρισης. Και είπατε γιατί δεν αφήνουμε τις εταιρείε ε, ήσυχε και ότι τις μπερδεύουμε με τους κανόνες. Σαν εποπτικοί φορείς δεν θέλουμε να τις αφήσουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να τις πρόχνουμε σωστή κατεύθυνση. Για τις κατευθυντήριες γραμμές εγκρίσεως πρέπει να αναθεωρηθούν οι προσανατολισμοί είναι μια υποχρέωση βάση νόμου βλέπετε. Και η νομοθεσία CRA 3 πρέπει να ληφθεί υπόψη για να αναθεωρήσουμε το πλαίσιο. Δεν μιλάμε για θέσπιση νέων νόμων, αλλά να ε, προσπαθήσουμε οι προσανατολισμοί να προσαρμοστούν στον κανονισμό. Για το δεύτερο, για τις μικρότερες εταιρείες αξιολόγησης Κάναμε προσπάθειες να δούμε τι προσέγγιση θα ακολουθήσουμε για να ενθαρρύνουμε ερχόμένες εταιρείε. να συμμορφωθούν με τους κανόνες. Για τα οικονομικά στοιχεία, τα δομημένα χρηματοστικά στοιχεία, είναι πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό για την αγορά. Θέμα το οποίο επεξεργαζόμεθα. Στα πλαίσια των απαιτήσεων STS. Και αυτό θα εισαχθεί στη διαδικασία του SCS. Και αυτό θα οδηγήσει σε μια βάση δεδομένων δημοσίας προσβάσεως για τα υποκείμενα στοιχεία που θα επιτρέψουν στους ενδιαφερομένους να προβούν στη δική τους ανάλυση, κάτι που είναι σημαντικότατο. Endorsement, Brexit, μελλοντικό μοντέλο. Έχω να πω το εξής για όλα αυτά. Για ρυθμιστικού λόγου θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιε αξιολογήσει. 72% των βαθμολογιών αυτών είναι από φορεί εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Η αναθεώρηση των προσανατολισμών για την έγκριση για το endorsement είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να διευκρινίσουμε κάποιε από τι εξουσίε τη ΕΣΜΑ όσον αφορά την εποπτεία των εγκεκριμένων βαθμολογιών αυτών, endorsed ratings. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι τρίτη χώρα μετά τον Brexit. Τα μεγαλύτερα ιδρύματα αξιολόγησης είναι στο Λονδίνο. Άρα είναι πολύ σημαντικοί οι κανόνες για το endorsement, για την εποπτεία. για το ERP μόλις ξεκίνησε αυτό πέρσι κατά την άποψή μας είναι πολύ ενδιαφέρουσα βάση δεδομένων πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα όταν ο κόσμος τα χρησιμοποιεί περισσότερο το σύστημα είναι πολύ πρόημο να ξέρουμε τι αντίκτυπο έχει το σύστημα αυτό το ERP για την αγορά ευχαριστώ η σύγκρουση συμφερόντων, το άλλο ερώτημα που ετέθη, έχετε να πείτε κάτι για τη σύγκρουση συμφερόντων. Um, όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, είναι από τις μεγάλες προτεραιότητες που έχουμε όσον αφορά την εποπτεία. Προσπάθησα να απαντήσω σε αυτό, στο πρώτο σημείο, που είπα πού εστιάζεται η ΕΣΜΑ ποιε προτεραιότητε. έχει. βλέποντας ε, τους ανεξάρτητους τα ανεξάρτητα διευθυντικά στελέχη, την όλη δομή, προσπαθούμε να μειώσουμε τα εφιστάμενα προβλήματα όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Διότι αυτό θα εμπόδιζε την ποιότητα των ε, βαθμολογιών της αξιολογήσεως. Στην ΕΣΜΑ κινούμεθα στα πλαίσια του επίπεδου 1 και του επίπεδου 2. Εντός της ανατεθής σας εντολής εξετάζουμε αυτά τα θέματα διακυβέρνησης και διαχείρισης. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε. Είναι σημαντικό η Επιτροπή μας να μπορεί να εξετάζει αυτές τις δύο εκθέσεις που αφορούν τους φορείς αξιολόγησης. Θα συνεχίσουμε από αυτού. Πάμε στο σημείο 11 της ημερησίας διατάξεως. Ο εισηγητής δεν είναι εδώ. Α, εσείς αντικαθιστάτε τον κύριο Τόιρερ. Μπορούμε να πάμε λοιπόν εκεί. Εξετάζουμε τις τροπολογίες. Γνωμοδοτήσεως για την Επιτροπή ΙΜΚΟ για τη διπλή φορολόγηση το Dispute Resolution Mechanism, το σύστημα διευθετήσης διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Βανούιτεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστεί ο εισηγητής όλους σας για την βοήθειά σας και για τις τροπολογίες. Πρόκειται για θέμα ευρύ συνένεσης ότι θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή των ε, φόρων για τις επιχειρήσεις ε, σε σχέση με τα κέρδη για τη διπλή φορολόγηση είναι βλαπτική. Ε, κάποιοι φορολογούμενοι προτιμούν την διπλή φορολόγηση παρά να μπλέουν σε διάφορες διαδικασίες που δεν παρέχουν για καμιά είδους ε, εγγύηση ε, για κάποια απόφαση που θα καταργήσει την διπλή φορολόγηση. Επομένω, με μεγάλη του χαρά είδε τι τροπολογίε τη σχετική ο εισηγητή, όπου τονίζεται ότι η επίλυση των σχετικών διαφορών θα πρέπει να γίνεται γρήγορα, με αποτελεσματικότητα και να έχει δεσμευτική ισχύ. Τονίζει στο κείμενό του ότι υπάρχει περιθώριο ούτω ώστε ο μηχανισμός πύλης διαφορών να διευρυνθεί και να είναι η διαδικασία πιο γρήγορη προτείνει συντομότερες, ε, μικρότερες προθεσμίες και κάπου μερικές αλλαγές στο περιφαρμογή και όταν ε, αποδεικνύεται ότι είναι επιτυχής ο μηχανισμός ε, τότε θα πρέπει να διευρυνθεί περισσότερο και να εφαρμόζεται σε όλες τις διαφορές σχετικές με διπλή φορολογία. Θεωρεί πάρα πολύ θετική αντίδρασή σας στις τροπολογίες και όπως είπαμε και πριν οι φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να εφίστανται την κύρωση, το πρόστιμο τέλο πάντων όσο κρατάει διαδικασία. Στι τροπολογίε επίση προτάθηκε ότι οποιοδήποτε φόρο που έχει αδίκω καταβληθεί θα πρέπει να επιστρέφεται. Αυτό ε, θα μπορούσε να είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει να διατυπωθεί και θετικά. Επίση θέλουμε να υπάρχουν μικρότερε προθεσμίε. Δεκτή η σχετική τροπολογία θα πρέπει να στο Κοινοβούλιο να είναι αποφασιστικό όποτε έχουμε τέτοιου είδους επαχθείς διαδικασίες υπερβολικές ε, σε διάφορα κράτη-μέλη. Οπότε έτσι έχουμε προστριβεί στην εσωτερική ε, αγορά. Και τόνισε ίδιο ο εισηγητής ότι αυτοί που έχουν οριστεί σε συμβουλευτικές επιτροπές και σε εναλλακτικές επιτροπές επίλυσης διαφορών θα πρέπει αυτοί να είναι ακέραιοι, να είναι αντικειμενική και αμερόληπτη. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια διαρκής επιτροπή που να εξασφαλίζει αυτό. Ε, με τέτοιο διαρκές όργανο θα πρέπει να οδηγήσει σε εύρυθμη διαδικασία και ταχεία και επίσης αυτός ο φορέας θα πρέπει να προσδίδει τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχουν τα μέλη αυτή της Επιτροπής. Και έτσι θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια στη διαδικασία, εν κατακλείδη ο εισηγητής και πάλι τονίζει το πόσο σημαντικό είναι το να είναι δίκαιο το σύστημα φορολόγηση των εταιριών και έτσι οι εταιρείε να μπορούν να ωφεληθούν πλήρω από την εσωτερική αγορά. Και βέβαια θεωρεί πάρα πολύ θετικό το υπάρχει ευρεία συνένεση ε, γύρω από ένα τέτοιο δίκαιο σύστημα. Σύντομα θα δίνουμε τις τροπολογίες για τις οποίες ε, ευχαριστεί, αλλά ευχαριστεί και τη γραμματεία μας για τη βοήθειά της. Ευχαριστώ πολύ. Επέστρεψε λοιπόν ο Πρόεδρος και έτσι θα του επιτρέψω να ξανακαθίσει την καρέκλα του, αλλά θα ζητήσω δύο λεπτά γιατί πρέπει και εγώ να γυρίσω στη δική μου θέση από όπου θέλω να λάβω το λόγο. So, next speaker. Επόμενη μιλήτρια, η Πέγμος Σπέχες. Όχι, ο Σάρλ πρώτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τι να πω, τι να πω, ύστερα από αυτήν την καταπληκτική παρουσίαση της Κούρεκ μέρους του Μιχαήλ Τόερερ. Ξεκινάμε μεγάλη επιτυχία η δουλειά μας. Τώρα περιμένουμε να δούμε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Απλώς θέλω να πω πως πιστεύω ότι με την έκθεση του έχει προχωρήσει προς την απόλυτα σωστή κατεύθυνση ο εισηγητής και βεβαίως χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιτάχυνση του μηχανισμού για τη διευθέτηση των διαφορών που προβλέπει. Τρία σημεία θέλω ιδιαίτερα να τονίσω πολύ σύντομα. Πρώτον, ε, σταθερή στήριξη της Επιτροπής διότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουν για χρόνια οι επιχειρήσεις να εκδοθεί απόφαση για διευθέτηση. Άρα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος του, της περικοπής των προθεσμιών. Επιτάχυνση επίσης μπορούμε να εξασφαλίσουμε εάν αυτή η Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται μέσα σε ρητές προθεσμίες και Μάλιστα αν είναι και μόνιμη η σύνθεση και η λειτουργία της περικόπτεται ακόμη περισσότερο ε, το διάστημα για τη διευθέτηση. Αυτός είναι ο κύριος στόχος και βεβαίως εξασφαλίζεται και μια ε, αίσθηση εμπιστοσύνης μεταξύ κρατικών αρχών, εάν είναι μόνιμη η σύνθεση. Η Συμβουλευτική Επιτροπή βέβαια δεν έχει ακόμα συσταθεί. Υπάρχει όμως η μόνιμη επιτροπή και ίσως μπορούμε με μια ε, δικαστική ε, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα χρειαζόταν πλέον μια δικαστική απόφαση για τον διορισμό μιας συμβουλευτικής επιτροπής. Άρα εξασφαλίστε και μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε σχέση με άλλα νομοθετήματα τώρα, οι ειδικέ τροπολογίε στόχο έχουν να συνδέσουν το θέμα αυτό με τα άλλα νομοθετήματα που ήδη υφίστανται. Ε, παραδείγματι, συμφωνία για διαιτησία ή διμερή συμφωνίε αποφυγή τη διπλή φορολογία στην οδηγία αυτή, ιδιαίτερα για την επίλυση των διαφορών, ε, ιδιαίτερα θέλουμε να τονίσουμε το πλεονέκτημα για τον φορολογούμενο και της φορολογικής έδρας αλλά και της ταχείας διαδικασίας. Ταυτόχρονα θα πρέπει σταδιακά όμως να προχωρήσουμε προς την κατάργηση της, ε, του νομοθετήματος για την ε, διαιτησία στη συγκεκριμένη υπόθεση για να διατηρηθεί ε, μια ενιαία κατάσταση. Επίσης, εάν έχουν ε, μια ένσταση απαράδεκτου από επιχείρηση ή φορολογούμενο, οι εθνικές αρχές μπορούν και να την απορρίψουν αλλά θα πρέπει να συμπληρώσουμε στο κείμενο ότι είναι υποχρεωτικός και υποχρεωτική και η έκθεση των λόγων, των αιτίων της απόρριψης στον φορολογούμενο για να μπορεί να καταλάβει γιατί απεριφθεί η ανστασία του. Κατά τα άλλα ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, ήταν πολύ καλό το σχέδιο εκθέσεως. Thank you. Ευχαριστώ. Περόν Περές για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, θα αντικαταστήσω την Ανλής Ντόντ. Uh, που δεν μπορεί να έρθει και θα διαβάσω αυτά που μου έγραψε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο που έκανε και τους άλλους συναδέλφους για την επικοδομητική προσέγγιση και τροπολογίες. Πολλές τροπολογίες εκθέσεως ε, είναι παρόμοιες και θα ενοποιηθούν μέσω συμβαστικών τροπολογιών που θα οδηγούν στη θέση του Κοινοβουλίου πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια καλή έκθεση Μα έδωσε μια καλή έκθεση η οποία θα βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφύγουν τις ζημίες που δημιουργούνται από τη διπλή φορολόγηση λόγω διαφορών των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά θα θέλαμε να δούμε πλήρη εφαρμοσμένη κοινή ενοποιημένη φορολόγηση των επιχειρήσεων που θα εμπόδιζε αυτού του είδους τα ζητήματα να προκύπτουν εμπρότης. Εν τω μεταξύ όμως αυτή η πρόταση θα επιτρέψει δημιουργία μεγάλη εμπιστοσύνη για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που θέλουν να λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση του εισηγητού βασίζεται στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μειώνει τον χρόνο που χρειάζονται οι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών για να επιλύσουν τι διαφορέ και φαίνεται ότι πολλοί συνάδελφοι μοιράζονται αυτή τη φιλοδοξία. Θα θέλαμε να μειωθεί το χρονοδιάγραμμα στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το ίμιση, ούτω ώστε να ευθυγραμμιστεί η διαδικασία με τον ετήσιο κύκλο επενδύσεων και επιχειρήσεων που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι αυτό ήταν το κίνητό τη για την πρόταση. Θέλουμε να μειώσουμε και το άκθος επί μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ίσως να πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το μηχανισμό ε, με την παρούσα πρόταση θα πρέπει να διερευνήσουν πιο το εθνικό δίκαιο και το εφαρμοστέα φορολόγηση στις δύο χώρες με τις οποίες έχουν διαφορά. Η πρόταση επίσης τις μικρές επιχειρήσεις ε, τις θέτει υπό χρονική πίεση για να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις αρμοδίων αρχών. Έχουμε υποβάλει τροπολογίες για να διορθωθεί αυτή η ανισορροπία και να υποχρεώσουμε τις αρμόδιες αρχές να ενημερώνουμε τους καταγγέλλοντες για δίποτε εξέλιξη, για δίποτε απόρριψη. Ισδήποτε αιτήσει για αύξηση του χρονοδιάγραμματος ή μείωση της διαφανείας δεν θα υποστηριχθεί από την ομάδα μας, διότι η μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια είναι βασικό στοιχείο για τη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας. Επίση, ζητούμε να γίνει αναθεώρηση οδηγίας και να συνδέεται με απόφαση του συνομοθέτου κατά πόσο θα πρέπει να εξακολουθεί να εφαρμόζεται ή όχι. Ελπίζουμε ότι μέχρι να γίνει αναθεώρηση θα έχουμε συμφωνήσει ένα πλήρες καθεστώς, οπότε ε, ίσως να μην χρειάζεται κάποιο στοιχείο αυτής της ε, πρότασης για κάποιες από τις μεγάλες εταιρείες τουλάχιστον. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και τους και εισηγητές για τις τροπολογίες που υπέβαλαν για την έκθεση και ελπίζουμε και προσβλέπουμε μάλλον στη συνέχιση της επικοδομητικής συνεργασία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος για το ECR. Πύρχον Βόρνερ Λένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η οδηγία που αφορά τη διπλή φορολόγηση και που ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι ένα κάτι που θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα στην εργασία. Θα έχουμε αύξηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και πρέπει να ε, ε, αυξάνονται οι φορολογικές ροές, χρειάζεται να έχουμε σαφέστατους κανόνες συνεπώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κάτι λειτουργικό, δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε όσον αφορά την ουσία του. Προτείνονται διάφορες τροποποίησεις. Οι τροποποίησεις θα οδηγήσουν σε πρόοδο. Θα πρέπει όμως η διαθέτηση των διαφορών να διέπεται από διαφάνεια να ρυθμίζονται οι διαφορές σε εύλογο χρονικό διάστημα για τις και για τις αρχές. Θα πρέπει η διαδικασία να οδηγεί σε βεβαιότητα και να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης για τις εμπλεκομένους φορείς. Ε, έχουν μειωθεί οι προθεσμίες που προβλέπονται και ίσως οι αυτές είναι πολύ ριζοσπαστικές για πολλούς λόγους αυτό ίσω δημιουργεί κινδύνους για τις επιχειρήσεις και για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι αρχές των κρατών μελών δεν έχουν απεριόριστους πόρου. υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών και η διαδικασία η οποία μπορεί να είναι πολύ γρήγορη σε ένα κράτος μέλο, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί σε άλλο κράτος μέλος. Δεύτερον, η εσωτερική εύξη της οικονομίας οδήγησε σε αύξηση της περιπλοκότητας των φατιθέσεων των διαφορών. Πιθανότατα νομικός και τεχνικός οι περίπλοκες περιπτώσεις δεν θα μειωθούν σε αριθμό. Αντιθέτως, εάν δεν κάνουμε σημαντική πρόοδο διοικητική, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα θετικά. Θα διαρκούν ε, επί πολύ οι διαδικασίες. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, πιο ανοιχτή προσέγγιση κυρίως όσον αφορά την επιλογή εμπειρογνωμόνων, η κοινοποίηση αυτών επίσης κάτι, είναι κάτι που πρέπει να ρυθμιστεί. Είδαμε το πώς κάποιοι, ε, η επιρροή των νομικών των επιφανών έχει αυξηθεί σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη μη ύπαρξη συγκρούσεων συμφερόντων κυρίως όσον αφορά την επιλογή των εμπειρογνωμόνων. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια. Η συγκέντρωση της εξουσίας θα πρέπει να αποκλείεται αν έχουμε μια επίκαιρη λίστα κατάλογο των εμπειρογνωμόνων. Αυτά και ευχαριστώ. Thank you for the e και τώρα για την Ευρωπαϊκή Νοτική Αριστερά. Ο <clears throat> κύριος Σουρμπάν Κρέσπο, ευχαριστώ πρόεδρε. Θεωρούμε ότι σήμερα όλες οι μεγάλες ε, εταιρείες ακολουθούν πρακτικές ε, διαφυγής ε, της φορολογικής βάσης και τιμολογική πολιτική ανάλογη τόσο να πληρώνουν φόρο σε κάποιες χώρες με λιγότερους φόρους και είναι λιγότερο από το 1% σε κάποιες χώρες ο εταιρικός φόρος. Άρα αυτοί που έχουν τα πολλά πληρώνουν τα πιο λίγα και είναι συνένοχοι σε αυτά τα κράτη γιατί ενεργούν προς το συμφέρον των, των και επίσης βάζουν τροχοπέδι στους ελεγκτές της εφορίας και αυτό είναι το πρόβλημα το φορολογικό στην Ευρώπη πως κάπτεται η κυριαρχία των ε, ε κρατών μελών και έτσι δυνατόν να υπάρξουν ε, υπηρεσίες από το δημόσιο τομέα ποιοτικές θα πρέπει μένω αυτό να είναι πρώτη προτεραιότητα για την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις. Δεν θα πρέπει να μας απασχολεί το αντίθετο του ορθού. Δηλαδή, ασήμαντες περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι η διπλή φορολόγηση, αλλά η διπλή αποφυγή. Γιατί για να καταπολεμηθεί το πρώτο σημαίνει ότι στην πραγματικότητα θα πρέπει να δούμε πόσο διευκολύνεται το δεύτερο. Αυτό μας απασχολεί. Και οπότε έτσι θα πρέπει να είναι πιο σύντομες οι η επιτάχυνση όλων των ε, φάσεων της διαδικασίας που συζητούμε και γι' αυτό είπαμε η, ε, η τριετής ε, προθεσμία για την ένσταση να είναι ενός έτους. Αυτό αρκεί. Άρα θα πρέπει να έχουν το χρόνο για να μελετήσουν την υπόθεση οι αρχές. Βέβαια πολλές φορές είναι περίπλοκες, άρα χρειάζεται κάποιο χρονικό περιθώριο στις κυβερνήσεις αλλά να μην παρελκύεται η διαδικασία και άρα θα πρέπει πριν να έχει υπάρξει η ένσταση του ενδιαφερομένου. Τώρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι ελεγκτές της εφορίας θα πρέπει να συμμετάχουν σε αυτές τις επιτροπές διαμεσολάβησης, επίλυσης διαφοράς, γιατί χρειάζονται τεχνικές γνώσεις που μόνο εκείνοι έχουν. Και έχουμε κατεβάσει μια τροπολόγια σχετικά με τον συνάδελφο Ουρτάσουν των Πρασίνων. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει δημοσιότητα των αποφάσεων σε όλες τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι το απόρριτο δεν στέκει εδώ όσον αφορά τη διεθνή φορολογία και είναι προς το γενικό συμφέρον η δημοσίευση της απόφασης να είναι πιο δίκαιες έτσι, οι αποφάσεις και θα πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι εφαρμόζονται οι νόμοι και χρειάζεται επομένως αυτή η διαφάνεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης δεν ε, συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι δηλαδή εάν υπάρχει κάποια προσφυγή στο αρμόδιο όργανο για την φορολόγηση θα πρέπει να αναστέλλονται οι συνέπειες της διαφοράς υποκρίσεων. Ε, αυτό επομένως ε, υποσκάπτει το έργο των αρχών και έτσι είναι δυνατόν καταχρηστικά να ασκούνται τα ένδικα μέσα αυτές οι ενστάσεις. Οπότε να αλλάξει αυτό το σημείο θέλω. Ευχαριστώ. Thank you for the Greens, Ernest Urtasun. Ernest Urtasun για τους πράσινους. Πρόεδρε, ευχαριστώ, όπως είπε και ο συνάδελφος. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ένα ισοδίκαιο φορολογικό σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και και αυτό το πιο σημαντικό από όλα είναι ο φόρος να εισπράτεται εκεί όπου ε, παράγεται το κέρδος. Σε αυτό θα επιμείνουμε, χρειάζεται οπωσδήποτε να CCTV σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι και η γραμμή των τροπολογιών μας. Είδαμε αρκετές τροπολογίες και από άλλους συναδέλφους που έχουν να κάνουν και με το χρονοδιάγραμμα, με την ένσταση, με το αίτημα για περαιτέρω ενημέρωση πληροφορία, για την εκκίνηση της διαδικασίας και την τελική απόφαση για τον φορολογούμενο. Προσπαθούμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις στην εργασία με τις άλλες ομάδες, αλλά θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα και τις διαφορετικές προτάσεις, ώστε η λύση στην οποία θα καταλήξουμε είναι καλύτερη και για τους επιχειρηματίες, αλλά και για τις αρχές. Και επίσης κύριο ζήτημα για μας. Ο προσδιορισμός ανεξάρτητων ε, ε, φορέων, αρμοδίων που θα προχωρήσουν στην επίλυση των διαφορών. Αυτή είναι ε, και η τροπολογία 156. Θέλουμε άτομα δηλαδή υψηλή ανεξαρτησίας με εγγυήσει ουδετερότητας που θα πρέπει σε ένα κατάλογο να κοινοποιούνται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο μηχανισμός, όπως τον προτείνει η Επιτροπή, ε, προβλέπει μία εξέριξη, το λέμε εμείς στην τροπολογία 166, η εγγύηση του έχει πολύ μεγάλη σημασία, το τονίζουμε στις τροπολογίες και η δημοσίευση της τελικής απόφασης επίσης είναι απαραίτητη για μας για να αποφεύγονται διαφορές με προσωπικό με μόνη απόκρυψη των προσωπικών στοιχείων ή των ε, στοιχείων που έχουν καθαρά προσωπικό χαρακτήρα. Ε, όλα τα άλλα στοιχεία πρέπει να δημοσιεύονται, δηλαδή τα σχετικά με την απόφαση. Κατά τα άλλα, θα συνεργαστούμε βέβαια με τον εισηγητή στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Η ευθυντή δεν είναι εδώ. Ενφ Κάπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση οδηγία για τη διαδικασία διευθέτησης ε, διαφορών διπλής φορολόγησης έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Έχουμε περίπου 900 ε, ε, διαφορές διπλής φορολόγησης στα δικαστηριά μας με πάνω από 10,5 εκατομμύρια ευρώ αντικείμενο που βρίσκονται σε εκκρεμότητα από το δικαστηρίων επί δύο και περισσότερα χρόνια. Χρειάζεται οπωσδήποτε περικοπή των ε, περιόδων ε, του, χρόνου που διαρκούν αυτές οι διαφορές ε, να διευθετούνται ταχύτερα και σε αυτό είναι σημαντική η πρόταση και θα πρέπει να κάνουμε επιτερετέρα προσπάθειες με τη συμβολή των εθνικών αρχών οι οποίες χρειάζονται καλύτερο υλικό, ανθρώπινο και λοιπό για να μπορούν να προχωρούν στη μελέτη της διαφοράς και την ολοκλήρωσή της, διαδικασίας της. Επίσης πολύ μεγάλη σημασία θα έχει η θέσπιση συμβουλευτικών επιτροπών είτε η σύγκληση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Αυτό και θα συντομεύσει τις διαδικασίες αλλά και θα βελτιώσει την ποιότητά τους. Είναι σημαντικό ε, οι ειδικοί που θα κληθούν όχι μόνο να είναι πραγματογνώμονες, να είναι ανεξάρτητοι, αλλά να μην είναι και μεροληπτικοί. Η αρχή της αποφυγής της διπλής φορολόγησης είναι ουσιώδης για την εσωτερική αγορά, για να λειτουργήσει καλά η εσωτερική αγορά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τα ταχύτερο δυνατό να βρούμε μια λύση. Και γι' αυτό περιμένω με αδημονία τις συμβαστικές τοπολογίες του εισηγητή. Ευχαριστώ. Δεν ζήτησε κανείς το λόγο στη διαδικασία Catch the Άρα να ξαναδώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Πού είναι. Α, δεν είναι εδώ. Uh, I can uh, read the which... διαβάσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 8 Ιουνίου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την πρωινή μας συνεδρίαση και θα ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας στις 3. Ευχαριστώ πολύ.